Allora se potete prendere posto per Μάλιστα, να σας καλωσορίσω λοιπόν στην Επιτροπή μας. Στην ε, ακρόαση αυτή θα ήθελα να καλωσορίσω ιδιαίτερα την Επίτροπο για την έρευνα, την καινοτομία και την επιστήμη. και τον εκπρόσωπο της Δανικής Προεδρίας από το Υπουργείο Επιστήμης. Θα τα ξεκινήσουμε και σήμερα το πρωί. Είχαμε κάποια προβλήματα με το χρόνο. Θα ήθελα λοιπόν να κάνετε ησυχία για να ξεκινήσουμε κατευθείαν. Το λέγω στην Ε. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε μέλη. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να ευχαριστήσω και την Επιτροπή Ήτρε που διοργάνωσε αυτή την ακρόαση για το πρόγραμμα Horizon 2020. Να ευχαριστήσω την Επιτροπή και τους εισηγητές ιδιαίτερα για τον χρόνο που έχουν αφιερώσει στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα να σας ε, διασ... Ναι, βεβαιώσω ότι έχετε την πλήρη υποστήριξη της Επιτροπής. Δεν υπάρχει λόγος να σας εξηγήσω στην παρούσα φάση τις λεπτομέρειες του προγράμματος. Παρουσίασα τις προτάσεις μας τον προηγούμενο Δεκέμβριο και έχει προηγηθεί γύρω ε, δύο γύροι ανταλλαγής ε, ε, απόψεων στην Επιτροπή τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο. Θα ήθελα ωστόσο να χρησιμοποιήσω την ευκαιρία αυτή για να κάνω κάποιες παρατηρήσεις σε ό,τι αφορά τις προτάσεις μας. Καταρχάς, συζητώντας ε, με διάφορους εμπλεκόμενους φορείς τους τελευταίους μήνες, ε, μου έκανε εντύπωση η συνένεση μεταξύ, έρευνα, μεταξύ των φορέων για την άποψη ότι είναι απαραίτητη η έρευνα και η επιστήμη για την οικοδόμηση ε, γέφυρας με πολλούς ε, κοινωνικούς τομείς. Επίσης υπάρχει κοινή αντίληψη ότι η φιλόδοξη πρόταση που έχουμε επιτάπητος μπορεί να μας βοηθήσει για να επιφέρουμε τις απαραίτητες αλλαγές που χρειαζόμαστε στην Ευρώπη. Σα σας υπενθυμίσω ότι το scoreboard που δημοσιεύθηκε τον περασμένο μήνα και το 2011 καταδεικνύουν ότι υπάρχει ε, μείωση της αύξησης Τη ανταγωνιστικότητα σε ό,τι αφορά την καινοτομία και ότι δεν κυφρέχουμε το χάσμα που υπάρχει με, τις, με την ε, Ιαπωνία, με την Κορέα. Και αυτό έγινε κυρίω στον ιδιωτικό τομέα. Κατά δεύτερον, παρά το γεγονό ε, ότι ήταν πολύ θετικέ οι πρώτε αντιδράσει για το πρόγραμμα Ορίζοντα 2020, ε, ξέρω ότι πολλά απομένουν να κάνουμε. Μπορεί να μην συμφωνούμε για όλε τι λεπτομέρειε. Ακούσαμε κάποια παραδείγματα σήμερα το πρωί από ό,τι άκουσα αλλά στην παρούσα φάση η συζήτηση στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο μας βοηθά να επικεντρωθούμε στους τομείς όπου χρειάζεται να υπάρχει καλύτερη διαλεύκανση, αν θέλετε, των βασικών αρχών του προγράμματος. Και στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να τονίσω ιδιαίτερα τη σημασία της ε, οικοδόμησης, της ε, ίδρυσης, αν θέλετε, συνεργειών με άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα προγράμματα συνοχής θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η αριστεία και η καινοτομία μπορούν να ανθίσουν σε όλους τους ε, ε, τομείς, σε όλες τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Και όπως αναφέρθηκε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει ένα τέτοιο έγγραφο για τους συνδέσμους αυτούς, τη σύνδεση αυτή μεταξύ του προγράμματος με τις πολιτικές συνοχές οι διάφοροι τομείς ε, της πολιτικής θα πρέπει να συνενωθούν για να αντιμετωπίσουμε τις μεγαλύτερες προκλήσεις στην κοινωνία και οι ερευνητές από διάφορους τομείς θα ενθαρρυνθούν να συνεργαστούν. Αυτό θα σημαίνει συνδέσμους μεταξύ των τριών πυλώνων του προγράμματος Ορίζοντας 2020, για παράδειγμα στον πυλώνα 1 για την αριστεία και την ε, επιστήμη θα μπορούσε να οδηγήσει στη χρήση νανοτεχνολογιών για την αντικατάσταση, για παράδειγμα, ε, των υφιστάμενων μέσων στα πλαίσια του δεύτερου πυλώνα. Και αυτά όλα θα μπορούσαν να περάσουν στον τρίτο πυλώνα. Στο θέμα της, του πολυτομιακού χαρακτήρα θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι οι κοινωνικές επιστήμες θα συμμετέχουν σε όλες αυτές τις κοινωνικές προκλήσεις πέρα από τις προκλήσεις που προσφέρονται για το ε, Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Συμβούλιο και αυτές οι νέες συνεργασίες δεν θα είναι πάντα εύκολες στην ίδρυσή τους αλλά ο αντίκτυπός του θα είναι τεράστιος κυρίες και κύριοι ανυπομονώ να συνεχιστούν οι καρποφόρες συζητήσεις στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο και το σημερινό η σημερινή εκδήλωση αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο. Είναι εξαιρετικό το έργο της κυρίας Μαντουρέλ, του κυρίου Έρελ, του κυρίου Σκίνου, του κυρίου Λάμπερτς και της κυρίας Ματίας. Σας καλώ λοιπόν όλους να κινηθείτε το συντομότερο δυνατόν προκειμένου να ολοκληρώσει την πρώτη ανάγνωση του το Κοινοβούλιο και να θέσει έτσι το πρώτο βήμα. Τέλος να πω δύο λόγια για κάποια βασικές πρωτοβουλίες που προβλέπονται τους επόμενους μήνε που είμαι βέβαιη ότι σας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Είμαι στη θέση να σας ανακοινώσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ε, υιοθετήσει μια ανακοίνωση μέχρι τα μέσα του 2012, η οποία και η ανακοίνωση αποτελεί αντίδραση στην έκκληση του Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου για να ολοκληρωθεί το αέρα μέχρι το 2014. Θα αναφέρει τα μέτρα που χρειάζονται για να πετύχουμε το σκοπό αυτό και θα επικεντρωθεί ιδιαίτερα στην κινητικότητα της σταδιοδρομίας και της κινητικότητας των επιστημόνων, της διασυνοριακής συνεργασίας, της κυκλοφορίας της γνώσης και της διεθνούς διάστασης της έρευνας. Κατά δεύτερον, η διεθνή συνεργασία στην έρευνα και στην ανάπτυξη θα ε, τύχουν ε, επεξεργασία σε ξεχωριστή ανακοίνωση μέχρι τα τέλη του έτους, καθώς το διεθνές προσκήνιο αλλάζει ταχαίω σε ό,τι αφορά την έρευνα και την ανάπτυξη και προσφέρει νέες προκλήσεις, νέες ευκαιρίες αλλά και νέες προκλήσεις, θα πρέπει να υιοθετήσει ένα νέο πλαίσιο συνεργασία η Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να δοθούν προτεραιότητες στις δραστηριότητε μας. Θα πρέπει να βελτιώσουμε τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020. Η ανακοίνωση αυτή θα θέσει ε, λεπτομερείς στόχους και κριτήρια και τις βασικές αργές λειτουργίες για την βελτίωση της ευρωπαϊκής δράσης στον τομέα αυτών. Και τρίτον, μέχρι τέλος του έτους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε μια επιτροπή θα ε, διαθέσει μια δεύτερη ε, αναθεώρηση, ενημέρωση των στόχων αυτών θα περιλαμβάνει τους δείκτες για την ε, νέα Ευρώπη του 2020 σύμφωνα και με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της, ε, του Φεβρουαρίου του 2011. Όπως ξέρετε, αυτά την χάνουν και υποστήριξη του ΩΣΑ και των στατιστικών υπηρεσιών. Τα πρώτα αποτελέσματα ελέγχονται στην παρούσα φάση. Και γι' αυτό λοιπόν είμαστε σε φάση προετοιμασίας του δίκτυ. Οι τρεις αυτές ανακοινώσεις που ανέφερα αποτελούν ε, μέρος του προγράμματος εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ε, ανακοινώθηκε πέρσι από το Σώμα των Επιτρόπων. Θα ήθελα να κλείσω λέγοντας, Πρόεδρε, ότι η θέση, η, ο ε, ορισμός προτεραιοτήτων σε ό,τι αφορά την έρευνα και την κοινοτομία αποτελεί προπόθεση για θέσει εργασία στο μέλλον. Και η πρώτερη εμπειρία μα καταδεικνύει ότι με τον τρόπο αυτό ε, θα μπορέσουμε με το βέλτιστο δυνατό τρόπο να εξέλθουμε τι κρίσει. γιατί χρειαζόμαστε Πρέπει να βγούμε από τη δυσχερή αυτή θέση, χωρίς όμως να ξεχνάμε ότι η, η Ευρώπη εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, εκπροσωπώντας 500, ε, 500 εκατομμύρια ε, πληθυσμό. Έχουμε ακόμα λοιπόν τεράστιο δυναμικό, ένα δυναμικό το οποίο θα πρέπει να πραγματοποιήσουμε με τη βοήθεια πρακτικών, αποτελεσματικών πολιτικών στην έρευνα και στην κοινοτομία και αυτό αφορά ακριβώς κυρίε και κύριοι το πρόγραμμα Horizon 2020. Ευχαριστούμε την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Επίτροπο και τώρα έχουμε τον ε, αρμόδιο Υπουργό εκ μέρους της Προεδρίας της δανέζική. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, φίλοι, πρώτα πρώτα επιτρέψτε μου να αρχίσω ευχαριστώντα το Κοινοβούλιο διότι εκάλεσε την Δανέζικη Προεδρία ε, σε αυτό το σεμινάριο για το ορίζον 2020 τώρα λοιπόν είναι η δική μου σειρά να σας πω πώς πάνε τα πράγματα, τι έγινε με τις διαπραγματεύσεις, να σας πω τις απόψεις του Συμβουλίου. Πιέζει ο χρόνος αν θέλουμε να καταλήξουμε ε, σε ε, κάποιο πρόγραμμα το οποίο να αρχίσει να τρέχει μέχρι το 2014 και μέχρι τώρα το Συμβούλιο πασχίζει ούτως ώστε να σημειωθεί συμφωνία μέχρι τα τέλη Μαΐου. Πιο συγκεκριμένα. Θέλουμε μια τέτοια προσέγγιση που να οδηγήσει σε συμφωνία ή στο Συμβούλιο επί της αρχιτεκτονικής του προγράμματος. Τώρα, για τα επιμέρους μέσα πολιτικής και υλοποίηση του προγράμματος αυτό θα συζητηθεί και θα συμφωνηθεί στη συνέχεια. Όλα αυτά θα γίνουν μόνο εάν εξασφαλίσουμε μια στέρη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γενικότερα και συγκεκριμένα με την Επιτροπή σας. Είμαι θα δε πεπισμένη ότι θα καταλήξουμε σε κάποιο πρόγραμμα το οποίο να είναι ευφυές και αποτελεσματικό. Βεβαίως και οι εμπλεκόμενοι έχουν απόψεις που μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Αυτό το, πώς να το λάβουμε υπόψη στην αρχή της διαδρομής και θα το λάβουμε μέχρι να ολοκληρωθούν διαπραγματεύσει. Τον περασμένο μήνα στην Κοπενχάγη οργανώσαμε μια υπουργική διάσκεψη. Συζητήθηκε το πρόγραμμα αυτό μεταξύ των υπουργών και των άλλων εμπλεκομένων. Ήταν ε, παραγωγικό αυτό ο διάλογο, είχαμε εκπροσώπου του επιχειρηματικού και του επιστημονικού κόσμου και είχε έρθει και η κυρία Καρβάλιο από το Κοινοβούλιο. Ήρθε και εξεπρο... εξεπροσώπησε συγγνώμη, την Επιτροπή σα. Τώρα, θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα βασικότερα σημεία. Για την αριστεία στην επιστήμη υπάρχει μια συνένεση να αποτελεί η αριστεία ένα βασικό κριτήριο και άλλωστε αυτό είναι προϋπόθεση για να είναι κανείς ανταγωνιστικός στην οικονομία. Επίσης, ε, αναφέρθηκε στη διάσκεψη ότι θα πρέπει να έχουμε λίγα μέσα πολιτικής για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Επίσης υπήρχε ευρεία συνένεση όσον αφορά τον προπολογισμό του Συμβουλίου ΑΕΡΣΥ. Και επίση τονίστηκε την σημαντική η κινητικότητα των νέων ερευνητών. Αλλά βέβαια θα πρέπει να δούμε και τα της σταδιοδρομίας τους. τονίστηκε πόσο σημαντική είναι η αριστεία ότι θα πρέπει να αντιληθούν πόροι από τα διαδοτικά ταμεία. Θα πρέπει ομένως, να υπάρχει μια συνέργεια και όλα αυτά τονίστηκαν επανειλημμένα στην Υπουργική Διάσκεψη. Θεωρήθηκε πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα όσον αφορά την, τον πρωτοπόρο ρόλο μας είπαμε ότι οπωσδήποτε θα πρέπει να είμαστε καινοτόμοι, θα πρέπει να συμμετάσχει ο ιδιωτικό τομέα ε, αναβαθμισμένα. Και επίσης θα τα καταφέρουμε εάν έχουμε στοχευμένα μέσα και απλούς κανόνες συμμετοχής. Επαναλαμβάνω ότι η απλούστευση είναι η ψήστη μας προτεραιότητα. Νέα ισορροπία να βρούμε μεταξύ εμπιστοσύνης και ελέγχου. Λιγότερη γραφειοκρατία. Αυτό το πνεύμα πρέπει να μας διαπνεί Συνεργασία επιχειρήσεων και πανεπιστημίων. Και αναφέρθηκε εδώ το βιομηχανικό δεκτορικό σε σχέση με αυτόν τον τομέα. Είπαμε ότι χρειάζεται η αριστεία, αλλά χρειάζονται και νέα προϊόντα στην αγορά. Πάρα πολύ βασικά όλα αυτά και έτσι θα πρέπει να από την παραγωγή και θα, όλα θα πρέπει να τα προωθήσουμε. Τώρα όσον αφορά το σημαντικό ζήτημα των ε, προκλήσεων που έχουμε θα πρέπει να προχωρούμε στοχευμένα. Χρειάζεται διεπιστημονική προσέγγιση, πολυκλαδική. Τονίστηκε και αυτό. Κοινωνικές επιστήμες ε, επίσης ε, παίζουν σημαντικό ρόλο και επομένως έτσι θα πρέπει να δούμε τις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Όταν λέμε για αλλαγή κλίματος, για την υγεία, για την ε, συμπεριφορά, όλα αυτά θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Επίσης, θα πρέπει να έχουν περιθώρια λιγμών οι ερευνητέ και να αναζητούν τις καλύτερες δυνατές λύσεις. Χρειάζεται ευελιξία και προσαρμοστικότητα για τους στόχους μας. Το ετώνησαν αυτό αρκετή στην διάσκεψη. Επομένω, ε, όλοι οι εμπλεκόμενοι, όπω ακούστηκε και το πρωί, άλλωστε είπαν ότι θα πρέπει να έχουμε πολυκλαδική προσέγγιση και διεπιστημονική. Να μην έχουμε κατάτμιση της προσέγγισης, αλλά να είναι σφαιρική. Επομένω, θέλουμε να καταλήξουμε για κάποια συμπεράσματα, όπω είπαμε μέχρι το τέλη Μαΐου στο Συμβουλίο. Και έτσι να συνεχιστεί ο διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και επίση θα έχουμε και εκείνο το σεμινάριο τη 8 η Μαΐου όσον αφορά τη χάραξη πολιτικής. Εδώ θα βάλω τελεία, Πρόεδρε, και έτσι θα ολοκληρώσουμε την εισήγησή μας. Κύριε Πέντερσεν, λέει η Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Και τώρα με μεγάλη μου χαρά σας παρουσιάζω τον ε, δόκτορα Λί. Προέρχεται από το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ για... και έχει την έδρα της καινοτομίας και γνωρίζει εις βάθος την κατάσταση στην Ευρώπη. Αλλά και στις ε, ΗΠΑ. Ποιος είμαστε στην Καλιφόρνια. 15 ε, χρόνια ασχολείται με από αυτές τις θέσεις με αυτά τα θέματα ο καθηγητής στατηγικό consulting παραχή δηλαδή συμβουλών είναι ερευνητή και σε Δουβλίνο, Βαρκελόνη, Βιέννη, Στουργάρδη έχει εργαστεί. Επομένως βλέπετε ότι έχει τεράστια εμπειρία και δεν περιορίζεται επομένω η δράση του στην Αμερική, στην Καλιφόρνια, στο Πανεπιστημίο. Έχετε τον λόγο, καθηγητά. Πρόεδρε Σαρτόρη, ευχαριστώ για την πολύ ευγενική εισαγωγή. Είναι μεγάλη τιμή να κάνω όλο το ταξίδι από την Silicon Valley στην καρδιά της Ευρώπης, στις Βρυξέλλες. Ήταν μακρύ το ταξίδι και ελπίζω ότι η μικρή ιστορία που θα σας πω θα είναι ενδιαφέρουσα και ίσως και λίγο διαφορετική από τις ε, υπόλοιπες που ακούσατε το πρωί. Να σας υπενθυμίσω ότι εγώ είμαι από τη πολιτεία της, τη Δημοκρατία της Καλιφόρνια και όχι από τη ΣΥΠΑ. Ε, έχουμε και τη Δημοκρατία του Τέξας, αλλά για αυτή δεν θα μιλήσω σήμερα. Η Καλιφόρνια είναι η, η έδρα του Silicon Valley Επίσης ε, θέλω να ευχαριστήσω την Κριστίνα Γκουτιέρες Κορτίνες. Αν δεν ήταν εκείνη δεν θα ήμουν εδώ. Και επίσης και ο Γκάι και η Σουζάνε ήταν πολύ χρήσιμοι γιατί με βοήθησαν να έρθω εδώ. Να πω κάποια πράγματα για μένα πολύ γρήγορα όμως για να επικεντρωθούμε στις τάσεις που επικρατούν στη Silicon Valley σήμερα. Θα μιλήσουμε για τον αντίκτυπο σαν βασική παράμετρο και του Horizon 2020 και την επιτυχία του και θα μιλήσουμε λίγο για την Ευρώπη, τι μπορεί να καταφέρει στο μέλλον, ε, ποια είναι η πραγματική ευρωπαϊκή κρίση, σε τι συνίσταται κατά τη γνώμη μου και συστάσεις. Θα μιλήσω για τον αντίκτυπο και όταν μιλάω για αντίκτυπο μιλάω για θέσεις εργασίας ως επιτοπλίστων. Αυτό είναι μια βασική παράμετρος για την επιτυχία του Horizon 2020. Τώρα, πώς κατανέμεται ο αντίκτυπος, πώς επιμερίζεται, ε, στα πλαίσια του προγράμματος πλαισίου του 2007 γιατί ήμουν ειδικό αξιολογητής τα τελευταία δύο χρόνια σε κανένα δύο περιπτώσεις και πολλά θέματα έχουν να κάνουν με την εμπορική εκμετάλλευση του προγράμματος του 2007 και θα παίξουν ρόλο και στο Horizon 2020 αν ληφθούν υπόψη κάποια, κάποια, κάποιες παράμετροι. Επίσης θα μιλήσω για την ανάλυση και αξιολόγηση του αντίκτυπου όπως κάνουμε στις Ηνωμένε Πολιτείες και τι σημαίνει αυτό όταν μιλάμε και για την ανάλυση του, 2000, του Horizon 2020 και να δούμε και την τάξη μεγέθους του αντίκτυπου του Horizon 2020 σε σχέση με τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Θα μιλήσω για τον αντίκτυπο γιατί αυτό σας ενδιαφέρει εσάς τους βουλευτές περισσότερο. Αυτό είναι σημαντικό γιατί συμβάλλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας και ενδιαφέρει στην περιοχή, στην εκλογική περιφέρεια, στη χώρα, την πατρίδα. Αυτό ενδιαφέρει πάρα πολύ και τους βουλευτές και τους δικούς μας και τους γερουσιαστές μας. Είναι το βασικό που τους απασχολεί. Οπότε θα πρέπει να δούμε πώς η έρευνα και η ε, καινοτομία μεταφράζονται σε θέσεις εργασίας, ποιότητα ζωής, ε, αυτά τα οποία κάνουν τη ζωή άξια να τη ζήσουμε. Θα μιλήσω και λίγο για τον μηχανολογικό σχεδιασμό, θα μιλήσω λίγο για χωνιά και αγωγούς, θα μπούμε σε κάποιες λεπτομέρειες. Έχω την τάση να είμαι πολύ ομός και ειλικρινής, καμιά φορά και προκλητικός για κάποιους από σας. Ε, θα σας δώσω κάποια στοιχεία λοιπόν για να... Και ελπίζω ότι θα σας ενδιαφέρουν αυτά εδώ στις Βρυξέλλες. Θα είναι μια διαφοροποίηση σε σχέση από αυτά που ακούτε συνήθως από άλλες πρωτεύουσες. Θα πάμε γρήγορα. Η κυρία Σαρτόρη ε, μίλησε για μένα. Εγώ είμαι από το, την, ε, όχι από τη ε, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, αλλά τη Σχολή Μηχανολόγων στο Στάνφορντ. έχετε ακούσει πάρα πολλά ονόματα επιχειρήσεων που έπαιξαν μεγάλο ρόλο και παίζουν ρόλο και κάνουν μεγάλη διαφορά και δημιουργούν και θέσεις εργασίας μεταξύ άλλων και καινοτομία και εδώ στην Ευρώπη. Η Σχολή Μηχανολόγων στο Στάνφορντ και σήμερα είναι στην καρδιά του οικοσυστήματος καινοτομιών της Silicon Valley. Να έρθετε να μας δείτε. Εγώ ε, στη Σχολή Μηχανολόγων διδάσκω καινοτομία και έχουμε σεμινάρια εβδομαδιαία. Ε, το τελευταίο ήταν στις 12 Μαρτίου όπου Φέραμε από την Silicon Valley και το San Francisco πολλούς ειδικού ε, επενδυτές, ε, καινοτόμους και ε, αυτοί που προσκαλέσαμε έχουν μεγάλη εμπειρία, έχουν δει το 70-80% των καινούριων επιχειρήσεων που ιδρύονται και τα τελευταία τέσσερα χρόνια που έκανα αυτό το σεμινάριο, το μεταπτυχιακό, ε, είδα πάρα πολλά ε, συστήματα, ε, την ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων. Είχαμε από την Ισλανδία μέχρι τη Ρωσία και τη Σκανδιναβία μέχρι το, τη Μεσόγειο. Καλύψαμε όλες τις περιφέρειες και ήταν πολύ ενδιαφέρον. Μέσα σε 10 εβδομάδες τα ε, τις καλύπτουμε αυτές τις περιοχές κάθε χρόνο. Ε, εγώ δεύτερη φορά προσκαλούμε να μιλήσω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρώτη φορά ήρθα πέρσι το Φεβρουάριο και συνάντησα και μέλη της Επιτροπής Βιομηχανίας ε, στα πλαίσια της ε, ειδική αξιολόγησης του προγράμματος πλαίσιο, οπότε μπόρεσα να δω λίγο από μέσα πώς τρέχουν τα προγράμματα της Ευρώπης γύρω από την έρευνα και την καινοτομία. Επίσης, ε, μια πολύ ενδιαφέρουσα προσωπική εμπειρία δική μου, που μου βοήθησε μεταξύ άλλων να καταλάβω το ευρωπαϊκό σύστημα και τι γίνεται εδώ, είναι όταν προσεκλήθη να γίνω ε, μέλος της Task Force για την έρευνα και την ανάπτυξη στην Ιρλανδία το 2009 και το 2010, γιατί έτσι κατάλαβα το Ιρλανδικό σύστημα και στην έρευνα και στα πανεπιστήμια και στις επιχειρήσεις και αυτό ήταν πολύ χρήσιμο πλαίσιο για να καταλάβω και άλλα συστήματα στην Ευρώπη με βάση το Ιρλανδικό. Επίσης τα τελευταία χρόνια ήμουν σύμβουλος σε ευρωπαϊκές νέες επιχειρήσεις που τώρα ιδρύονταν σε διάφορες περιοχές, διάφορες επιχειρήσεις. Η Ντέμλερ στη Στουτγάρδη χρηματοδοτούσε το πρόγραμμα και έτσι ε, γνωρίζω θέματα που αφορούν τον κλάδο το, της μηχανολογίας. Επίσης ε, ήθελα να εξετάσω και έκανα μελέτη διαφόρων πτυχών του Horizon 2020 προετοιμάζοντας την ομιλία μου. Ε, για να δούμε λοιπόν τώρα τη Silicon Valley. Όσοι δεν έχετε πάει, είναι μικρή περιοχή πρέπει να πω. Είναι λίγο κάτω από 3 εκατομμύρια οι κάτοικοι, 1,3 ε, εκατομμύρια θέσει εργασία. Ε, Υπάρχει λογισμικό, ποιοι είναι οι τομείς ανάπτυξη, δηλαδή ενέργεια, βιομηχανία, μέσα, ψυχαγωγία, βιοτεχνολογία, 40% του επιχειρηματικού κεφαλαίου τον ΗΠΑ συγκεντρώνεται εκεί. Τώρα τα κινητά και το cloud οι ε, ε, τώρα αναπτύσσονται πάρα πολύ, εκρηκτική θα λέγαμε η ανάπτυξη. Επίσης έχουμε το Android της Google, iOS της Apple, Windows, Microsoft, ε, το Windows, Windows Nokia αυτή η εταιρική σχέση τώρα αυξάνεται πολύ ε, είναι μια ολόκληρη οικονομία που αναπτύσσεται πολύ ταχύτερα στην Silicon Valley από ότι στην υπόλοιπη ε, βιομηχανία. Επίσης είπα ότι τώρα έχουμε μια συγχώνευση mobile και cloud ε, το mobile και cloud συγχωνεύεται γύρω από την ψηφιακή φροντίδα για την υγεία, αυτό τομέα, και πολύ επιχειρηματικό κεφάλαιο και έρευνα διοχετεύονται εκεί για να ε, αναπτυχθούν τα καινούργια σύγχρονα συστήματα, τα ψηφιακά συστήματα φροντίδας για την υγεία. Αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον για σας είναι μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε το Φεβρουάριο και που επικεντρώνεται στην δημιουργία θέσεων εργασίας ε, αυτό που λέμε οικονομία app που τι σημαίνει. Σημαίνει ανάπτυξη λογισμικού γύρω από τα ε, Apple, Android, Rims, BlackBerry και Nokia και Nokia Microsoft και πολλοί ε, συμμετείχαν στη μελέτη και είδαν ότι περίπου μισό εκατομμύριο θέσεις εργασίας μπορούν να διατηρηθούν ή να δημιουργηθούν μέσα σε τέσσερα χρόνια, το τονίζω αυτό, γύρω από τις apps. Οπότε αυτό είναι νέο μέτρο συγκριτικής αξιολόγησης και για τη ΣΥΠΑ και διεθνώς. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ σοβαρή πρόκληση αυτό και για την Ευρώπη και για οποιαδήποτε άλλη περιοχή που μπορεί να μην υπογράμμισε και να ανέδειξε το λογισμικό και τα έξυπνα τηλέφωνα, smartphones, mobile, cloud όπως είπα και η Silicon Valley συγκεκριμένα. Οπότε το βασικό είναι 500.000 θέσεις εργασίας σε τέσσερα χρόνια, όχι μόνο στη Silicon Valley, σε όλη την ε, Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ως επιτοπλίστων στη Silicon Valley όμως. Είναι ένας τομέας λοιπόν που βλέπουμε η ΕΠΑ και η Silicon Valley να ξεχωρίζει από άλλα σημεία του κόσμου, γιατί πραγματικά έχουμε πολύ δυναμικότερη ανάπτυξη και επιτάχυνση της ανάπτυξης που δεν φαίνεται σε πιο παραδοσιακούς τομείς όπως ιατρικά μηχανήματα, ημιαγωγούς κλπ. Αυτά είναι ε, γύρω από το ε, ε, Venture Capital Angel Network κλπ. Και είναι πολύ σημαντική η συμμετοχή στην οικονομία UP. Πολύ σύντομα τώρα ένα σημείο τεσ, αναφοράς τεσσάρων ετών Έχουμε τώρα ε, ένα γράφημα από το 2002 το 2011 και εδώ έχουμε ανατομέα τι είναι πολύ σημαντικό στα πλαίσια της οικονομίας ΑΠ. Από αριστερά βλέπουμε το μεγαλύτερο κομμάτι που είναι κόκκινο και που είναι το διαδίκτυο και το λογισμικό του και μετά φέρονται και οι υπόλοιποι το θα τα δείτε γιατί είναι, ε, τα έχω και ε, ετοιμάσει για σας. Ε, ας δούμε λοιπόν τώρα τι αντίκτυπο έχει η Silicon Valley στην Ευρώπη. Πάμε σε τρεις τομείς στα πλαίσια του αντίκτυπου. Καταρχήν είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι μεγάλες πρόοδοι και άλματα έγιναν γύρω από την, τα προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης της Κομισιόν τα τελευταία χρόνια και χαίρομαι πολύ γιατί το Horizon 2020 ε, τώρα σαφώς στοχεύει στο να ξεπεράσει ε, κάποια προβλήματα που είχε το πρόγραμμα πλαίσιο 7 τα οποία είχα εντοπίσει και εγώ επειδή ήμουν ε, ειδικό αξιολογητής ε, σε συνεδρίες αξιολόγησης από ειδικού που άκουγα του εκπροσώπους τη Κομισιόν να μου λένε να μην θεωρήσω την εμπορική εκμετάλλευση ω κομμάτι του αντίκτυπου και αυτό αρνήθηκα εγώ βέβαια να το κάνω και δεν συμφώνησα γιατί δεν νομίζω ότι έτσι ε, προσφέρουν υπηρεσίες στους λαού τη Ευρώπη. Πολύ πρόοδος έγινε στο μοντέλο του και την εφαρμογή του Horizon 2020 σε σχέση με το FP7, το πρόγραμμα πλαίσιο, και γύρω από την Ένωση της Καινοτομίας, εσείς τα ξέρετε καλύτερα, τα ενιαία αυτά ε, συστήματα ε, διπλωμάτων έβρεση τεχνίας, ε, αυτά είναι θέματα τα οποία προχωρούν στην Ευρώπη. Εγώ θα μιλήσω για τη διασυνοριακή επένδυση ένα επιμέρους στοιχείο που προέκυψε και από τη δικιά μου τη συμμετοχή στο Task Force της Ιρλανδίας για την καινοτομία είναι ότι πρώτη φορά συμπεριλήφθη ο σχεδιασμός προϊόντων ως κομμάτι της στρατηγικής καινοτομίας της Ιρλανδίας γιατί αυτό το στοιχείο έλειπε και στη Σχολή Μηχανολογίας και στις ιατρικές. Τώρα έχουμε συνεργασία με δύο Ιρλανδικά πανεπιστήμια από το Στάνφορντ για να έχουμε ε, βελτίωση όλων αυτών στα Ιρλανδικά πανεπιστήμια και πιστεύω ότι μπορούμε έτσι να αναβαθμίσουμε το σχεδιασμό στα πλαίσια της ατζέντα καινοτομία της Ευρώπης. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό καινούριο στοιχείο. Θα μιλήσουμε και για την κατανομή, ε, τον καταμερισμό του αντίκτυπου στα πλαίσια του Horizon 2020. Ε, πολύ σημαντικό είναι να δούμε το στοιχείο των νέων εταιριών και την εμπορική εκμετάλλευση. Ε, επίσης εδώ έχουμε τις ε, βασικές εστίες της Ευρώπης στα πλαίσια του, του προγράμματος 2012 της Ευρώπης του 2012, ίσως κάποιες δεν έχω συμπεριλάβει κάποια σημεία πολύ σημαντικά ε, πάντως έχουμε το Λονδίνο, Ελσίνκι, είναι πολύ σημαντικά στην επιχειρηματικότητα. Η Ζηρίχη, η Στοκχόλμη, το Δουβλίνο επίσης αυξάνεται και στην επιχειρηματικότητα, στη σημασία του και στο επιχειρηματικό κεφάλαιο. Οπότε ο χάρτης αυτός ε, προειδάζει για τον επόμενο χάρτη, γιατί αν το έχετε υπόψη σας, ε, που αναπτύσσεται κυρίω η επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη τα επόμενα 5-10 χρόνια, τι θα συμβεί με τις νέες εταιρείε που μπορεί να δημιουργηθούν από το FP7 και από το Horizon 2020. Προς τα που θα κινηθούν οι νέες εταιρείες ούτως ώστε να έχουν επιχειρηματικό κεφάλαιο, να έχουν ε, ε επιταχυντές κλπ. Αν δεν υπάρξει αλλαγή, στην ε, κατανομή του επιχειρηματικού κεφαλαίου, οι νέε εταιρείε από την Ανατολική Ευρώπη και από τη Μεσόγειο θα πάνε αλλού για να βρουν πρόσβαση σε επιχειρηματικό κεφάλαιο, για παράδειγμα. Και ο κίνδυνο εδώ είναι ότι μπορεί να υπάρξει τελείω άνηση κατανομή των ωφελιών και του αντίκτυπου τη εμπορική εκμετάλλευση του Horizon 2020 και αυτό στο τέλο θα γίνει πρόβλημα πολιτικό στου κόλπους τη Ευρωπαϊκή Ένωση αν δεν αντιμετωπιστεί. Εδώ λοιπόν χρειάζεται επένδυση διασυνοριακά και αυτή είναι μια πρωτοβουλία η οποία γίνεται από την Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων, ε, DG Enterprise, και νομίζω ότι θα πρέπει να συνδεθεί ε, με τρόπο ε, καλό, σωστό, στο πρόγραμμα Horizon 2020, γιατί μπορεί να επηρεάσει την ίση η μίση κατανομή των θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν, των εμπορικών ε, αξιοποιήσεων των προγραμμάτων από το Horizon 2020. Έτσι λοιπόν ε, θα πρέπει να βρεθούν κατάλληλοι επενδυτές. Αυτή είναι μια διαδικασία που συνεχίζεται. Θα υπάρξουν πορίσματα τον Ιούνιο γιατί εξετάζονται όλα αυτά υπό την ε, προεδρία του Άντωνη Κλάρκ. Αυτά για την κατανομή, λοιπόν, τον καταμερισμό του αντίκτυπου. Τώρα θα μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες, ανάλυση και αξιολόγηση του αντίκτυπου και την προσέγγιση που έχουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες που είναι από κάτω προς τα πάνω. Και εδώ πάμε στα, στη θεωρία με, με το χωνί και τους αγωγούς. Χρησιμοποιούμε χωνί και αγωγό για να δούμε πώς ε, παίρνουμε τις ε, εταιρείε που πρώτο ιδρύονται μέσα από τα διάφορα στάδια ή τεχνολογίες από την ιδέα μέχρι το προϊόν και ποια είναι τα ποσοστά θνησιμότητας ή αποτυχία στα διάφορα στάδια. Και αυτό είναι ε, κάτι που το κάνουν όλοι οι επενδυτές και τους απασχολεί πάντοτε. Εδώ έχουμε τον αγωγό της ε, καινοτομίας ε, από ε, την Ιρλανδία ε, και την ε, έκθεση του Task Force. Βλέπετε εδώ σχηματικά τον αγωγό που δημιουργήσαμε για την Ιρλανδία. Ένα παράδειγμα, έχουμε τις ιδέες στην αρχή, τα μοντέλα που οδηγούν σε ίδρυση επιχειρήσεων και περνάνε από διάφορα βήματα μέχρι την έξοδο. Έξοδο σημαίνει πώληση και επιστροφή στην αγορά εργασίας. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Ε, δεν έχουμε, ε, έχουμε εξελίξεις, πωλήσει εταιριών και δεν παγώνουν οι μικρές εταιρείες χωρίς να δίνουν αποτελέσματα. Ε, αυτή είναι η πολιτική καινοτομιών που παρουσιάζεται με, αυτό, με αυτούς τους αγωγούς. Επίσης, αυτό χρησιμοποιούμε όταν έχουμε υπόψη μας τις νέες εταιρείες ε, τη τεχνολογίας. έχουμε εδώ το πρώτο στάδιο ε, από τα σπάργανα δηλαδή, ε, από πανεπιστήμια, από κονσόρτσια σε άλλους ε, χώρους που περνάνε από τη διαδικασία του αγωγού, διάφορα στάδια, σχηματικά δηλαδή από το 1 μέχρι το 4 στάδιο και σε κάθε στάδιο κάποιες εταιρείε αποτυγχάνουν για τον α ή β λόγο. Οι περισσότερες αποτυχίες είναι στο πρώτο στάδιο ανάλογα όμως και με τον τομέα και τη χώρα. Μπορεί και μέχρι 90% των εταιριών να αποτύχουν. Έχουμε λοιπόν αριστερά το, τις εισρωές, πολλές αποτυγχάνουν και στο τέλος δεξιά έχουμε τις επιτυχημένες που είτε αγοράζονται είτε πολλούνται κλπ. Exit δηλαδή έξοδος. Έχουμε τα ποσοστά αποτυχίας ε, τα οποία τα γνωρίζουν οι επενδυτές ε, και τα παρακολουθούν σε κάθε χώρα γιατί έτσι θέλουν να κρίνουν και να αποφασίσουν πού θα επενδύσουν, πού βρίσκονται, ε, πόσες εταιρείες είναι σε ποια ε, σε ποιο στάδιο. Οπότε αυτά είναι πραγματική ζωή δεδομένα ρεαλιστικά που χρησιμοποιούνται για να κατασκευαστούν οι αγωνοί. Πάλι η προσέγγιση είναι από κάτω προ τα πάνω και οι κυβερνητικέ ε, ε, υπηρεσίε το χρησιμοποιούν αυτό το μοντέλο. Όταν προγραμματίζουμε ένα πρόγραμμα, αναπτύξουμε μια αίσθηση του πόσε επιτυχεί εταιρείε θα έχουμε στο τέλος. Μπορούμε μετά να το βάλουμε αυτό, να χρησιμοποιήσουμε ένα πολλαπλασιαστή, θα το δούμε αυτό, και να καταλήξουμε στις ε, θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν. Και το Ίδρυμα Επιστημών το χρησιμοποιεί ε, για τις νέες εταιρείε ε, να κρίνει τη διαδικασία τους, το μέλλον τους την, ε, τις φάσεις ανάπτυξής τους και αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στο Horizon 2020. Ε, ε, ε, ίσως αυτή είναι η μοναδική εξίσωση που θα δείτε σήμερα, ε, για να μην σας κουράσω. Η σημασία της ανάλυσης του αγωγού είναι μια ε, προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω που χρησιμοποιείται και από τους επενδυτές και τους πολιτικούς όμως όταν κρίνονται προγράμματα ε, υποστήριξης των επιχειρήσεων. Γιατί έτσι βλέπουμε τις διάφορες φάσεις ανάπτυξης από όπου περνάνε οι επιχειρήσεις. Ε, και το βασικό εδώ είναι το ποσοστό αποτυχία σε κάθε στάδιο. Για παράδειγμα, στην περίπτωση της Ευρώπης μπορεί να αναπτύξει κανείς ανάλυση με βάση το χωνί για κάθε χώρα στην Ευρώπη με βάση δεδομένα από τον τομέα των νέων επιχειρήσεων που ιδρύονται. Κάποιες χώρες μπορεί να δυσκολευτούν περισσότερο γιατί δεν έχουν αρκετά στατιστικά στοιχεία και στατιστικούς που θα τα επεξεργαστούν, αλλά μπορεί να είναι ενδιαφέρον αυτό το στοιχείο για την πολιτική καινοτομιών και σε εθνικό επίπεδο. Γιατί θα αρχίσει κανεί να παρακολουθεί τι εταιρείε ε, που περνάνε από τον αγωγό, θα αξιολογεί τα ποσοστά και θα μετράει τα ποσοστά αποτυχία για να ξέρει που βρίσκεται στο χωνί τη καινοτομία, στον αγωγό τη καινοτομία και να δει τι θα κάνει για να βελτιώσει τα ποσοστά αποτυχία και να ενισχύσει τις επιτυχημένες καινούργιες εταιρείες. Αυτό μπορεί να λειτουργήσει σε όλη την Ευρώπη. Επίσης μπορούμε να έχουμε ανατομέα αξιολόγηση για τα ποσοστά αποτυχιών. Αν δούμε δηλαδή τους διάφορους τομείς μπορεί να είναι άλλα και τα ποσοστά αποτυχίες. Μπορεί στα ιατρικά μηχανήματα να είναι διαφορετικά τα ποσοστά αποτυχίες από ό,τι στην, ε, στις τεχνολογίες ε, πληροφορίας και επικοινωνίας προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω, όπως σας είπα, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος της θέσης εργασίας του Horizon 2020 ε, με την προϋπόθεση ότι έχουμε μεγάλο αριθμό προγραμμάτων για να το κάνουμε αυτό και να έχουμε και ιστορικά δεδομένα. Δηλαδή τι προέκυψε από τα προγράμματα και τα έργα του FP7, του προγράμματος πλαίσιο 7. Είναι χρήσιμο αυτό για να αναλύσουμε τον αντίκτυπο και στο μέλλον. Ε, πάνω στη βάση των συνομιλιών που είχα τις τελευταίες ημέρες και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατάλαβα ότι το FP7 δεν χρησιμοποίησε πολλές τέτοιου είδου αναλύσει. διορθώστε με αν κάνω λάθο, αλλά έχω την εντύπωση ότι η Γενική Διεύθυνση ε, της Έρευνας δεν, χρησιμοποιεί, ε, δεν χρησιμοποίησε την ανάλυση των ε, αγωγών για να αναλύσει το FP7 και το Horizon 2020. Έχω την εντύπωση ότι οι αριθμοί των θέσεων εργασία που συσχετίζονται με, την, ε, με τον κατάντι οικονομικό αντίκτυπο του Horizon 2020 βασίζονται μάλλον σε μακροοικονομικά μοντέλα. Δεν γνωρίζω πολύ καλά από πού παίρνουν δεδομένα αυτά τα μοντέλα, δηλαδή πάνω σε ποιες υποθέσεις εργασίας βασίζονται. Ε, περνάμε στο επόμενο θέμα, ε, που είναι η τάξη μεγέθους του αντίκτυπου για τη δημιουργία νέων θέσεων στο Horizon 2020. Έχει αναφερθεί ότι η εκτίμηση του αντίκτυπου, μόνο εκτιμήσεις είναι αυτές, είναι ότι μέχρι το 2025 περίπου 3,7 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας θα μπορούσαν να δημιουργηθούν από το Horizon 2020, δηλαδή μέσα σε 10 χρόνια, 12 χρόνια. Συγγνώμη. <clears throat> Αν δούμε τη δεξιά πλευρά της διαφάνειας θα δούμε 7,5 ε, κουτάκια που το κάθε ένα χρησιμοποιεί ε, αντιπροσωπεύει 500.000 θέσεις εργασίας που χρησιμοποιούνται από τις οικονομίες app. Αν πάρουμε αυτό ως ε, μέτρο συγκριτικής αξιολόγησης μπορούμε να δούμε πόσες θέσεις εργασίας θα χρησιμοποιηθούν μέσα σε ένα χρονικό διάστημα. Αυτό το 3,7 μέσα σε 12 χρόνια, 3,7 εκατομμύρια δηλαδή θέσεις εργασίας και σημαίνει ότι στα πλαίσια του Horizon 20 θα είναι διπλάσιος ο ρυθμός δημιουργίας θέσεων εργασίας από την οικονομία ΑΠ στι Ηνωμένες Πολιτείες με λιγότερες από τις μισές επενδύσεις στις ε, τεχνολογίες ε, ε, πληροφορίας και ε, επικοινωνία στο ICT. Έτσι λοιπόν, ε, με βάση την ανάπτυξη στη ΣΥΠΑ, γύρω από το λογισμικό σε επιτοπλίστων, που είναι ο, ο ραγδαία αναπτυσσόμενο τεχνολογικός τομέας, τα 3,7 εκατομμύρια στα 12 χρόνια είναι πραγματικά απίστευτο αριθμό. Και αν αυτό το αναγάγουμε στο προηγούμενο κομμάτι που κάναμε την ανάλυση από κάτω προ τα πάνω, θα έλεγε, ε, η ερώτηση είναι μια ανάλυση από κάτω προς τα πάνω ε, και η ανάλυση με τους αγωγούς που δείξαν πριν θα υποστήριζε τον αριθμό των 3,7 εκατομμυρίων εσθέσεις. Το μέλλον τώρα. Ε, θεωρώ ότι η ευρωπαϊκή κρίση δεν αφορά το ευρώ ούτε τα, ε, το εθνικό χρέος αλλά είναι μια κρίση καινοτομίας αφορά τις σημερινές προκλήσεις και δυστυχώς αυτό δεν το προσέχουν πολύ ούτε τα ΜΜΕ ούτε το κοινό. Δεν, έχει, δεν το έχουν καταλάβει, δεν τους το εξήγησε κανείς καλά τι είναι η κρίση. Με την κρίση καινοτομία τι εννοώ. Όλα αυτά έχουν να κάνουν βέβαια και με τη Silicon Valley που έχει το μεγαλύτερο ρυθμό χρηματοδότηση δημιουργία θέσεων εργασία, δημιουργία επιχειρήσεων κλπ. Όλα είναι σχετικά βέβαια αυτά που λέω και γι' αυτό λέω ότι ίσω ακουστώ και προκλητικό σε κάποια αυτιά δικά από τη Silicon Valley εμείς βλέπουμε ότι η Ευρώπη πάσει από χρόνια απουσία ε, συνεχιζόμενης και επιταχυνόμενης δημιουργίας θέσεων εργασίας, απουσία ε, νέας, νέων γενεών καινούριων εταιριών που θα προέρχονται από εταιρείες στον τομέα της τεχνολογίας, πληροφορίας και επικοινωνίας που θα πάνε στο χρηματιστήριο να εισαχθούν ή που θα αγοραστούν και που παρουσιάζονται στο Google και την ολόκληρη γενναία, το ίδιο και στο, Facebook, στο Facebook. Συγγνώμη. Ε, θα υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείε ε, που θα εμφανίζονται εκεί. Αυτό είναι ένα φαινόμενο καταράκτη το, για την ε, ορατότητα αλλά και την ανάπτυξη των καινούριων, των, νέων των εταιριών που νέο δημιουργούνται. Ε, στην Ευρώπη αυτό δεν υπάρχει τόσο πολύ. Στην Αμερική παρουσιάζεται αυτό το φαινόμενο, ε, υπάρχουν δηλαδή ε, και είναι πολύ πιο ορατές σε πολλά επίπεδα. Δεν υπάρχει επίσης μια υποδομή για την ταχεία αναβάθμιση των ευρωπαϊκών τεχνολογιών. Επίσης δεν υπάρχουν πάρα πολλά καινούρια προϊόντα προκλητικά που ταράζουν τα νερά και αλλάζουν τον ρούν των πραγμάτων στην Ευρώπη. Ε, ίσως ε, το θέμα του λογισμικού δεν το ε, έχει συνειδητοποιήσει η Ευρώπη όσο οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Silicon Valley ως μια βασική συνιστόσα για την καινοτομία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. υπάρχουν εταιρείε που θα μπορούσαν όμως να συμβάλλουν όταν δεν επικεντρωνόμαστε στο λογισμικό, όταν ε, πάμε στους παραδοσιακούς ε, τομείς ε, καινοτομίας, ε, ας πούμε συστήματα μαζικής μεταφοράς, εδώ ξεπερνούν οι Ευρωπαίοι τους Αμερικανούς. Το θέμα όμως είναι ότι οι πολλαπλασιαστές σε αυτούς τους παραδοσιακούς τομείς είναι πολύ χαμηλότεροι από ό,τι στο λογισμικό. Οπότε, αν καλλιεργήσετε το λογισμικό, ε, θα έχετε κέρδος οι Φιλανδοί. Δεν έχουν κάνει πίσω, ούτε θα πρέπει να πείτε ε, ή το ότι α, δεν μπορούμε να φτάσουμε τις Ηνωμένε Πολιτείε. Ε, δεν πρέπει να φύγουν οι επιχειρήσεις ε, που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν στην Ευρώπη και να έρθουν στην ΕΠΑ, στη ΗΠΑ. Ε, δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει μια Silicon Valley στην Ευρώπη. Ε, ε, υπάρχουν τομείς ε, και στη ΣΥΠΑ που είναι πολύ πιο πίσω σε σχέση με το λογισμικό και έχουν πρόβλημα εκεί η αυτοκινητοβιομηχανία ή κάποιες μεγάλες επιχειρήσεις ε, στις μεσοδυτικές πολιτείες πάντως παρατηρείται ότι εκεί που το software δεν έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ είναι και λιγότερες οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται. Καμιά φορά δεν μπορούμε να εξαρτώμεθα στα ερευνητικά ιδρύματα και στην Ευρώπη ισχύει αυτό πολύ. Δεν μπορεί κανείς να περιμένει από τα ερευνητικά ιδρύματα <clears throat> να κάνουν τη διαφορά και να κινούν τα νήματα, εννοώ δηλαδή να ε, βοηθούν την ανάπτυξη των εταιριών ή να ε, ε, συμβάλλουν και να προωθούν την εμπορική εκμετάλλευση. Ε, ακούσαμε και σήμερα το πρωί ότι η επιστημονική αριστεία είναι ο πρωταρχικός του στόχος. Εμείς πιστεύουμε ότι μπορούμε αυτή την αριστεία και την καινοτομία μπορούμε να τα συγκεράσουμε στο ίδιο ίδρυμα. Εδώ στην Ευρώπη είναι πιο ξέχωρα αυτά τα πράγματα και στα πανεπιστήμια και στα ερευνητικά ιδρύματα. Το στοιχείο της καινοτομία ε, μπορεί να ενσωματωθεί στο στοιχείο της ε, ε, επιστήμης βασικής έρευνας. Έτσι θα υπάρχουν φορείς που θα έχουν σχέση με την αγορά και θα βοηθήσουν να γίνει πιο καινοτόμος ο επιχειρηματικός κόσμος. Επίσης είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι η έρευνα δεν είναι η μόνη κινητήρια δύναμη για την καινοτομία. Έγινε εδώ ένα σημαντικό σφάλμα, το οποίο παρατηρήσαμε και στην Ιρλανδία, γιατί το Task Force στην Ιρλανδία ήταν γύρω από τα πανεπιστήμια και την καινοτομία και εκτός από μερικές σελίδες που τις βάλαμε εκεί πέρα για να μην δημιουργηθεί η αμηχανία στον Πρωθυπουργό, ε, λίγα πράγματα είπαμε για την καινοτομία των επιχειρήσεων. Αυτό είναι ένας τομέας όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να τον προωθήσει, να το μελετήσει γιατί η καινοτομία με βάση την έρευνα δεν αρκεί για να δημιουργήσει θέσεις εργασίας μακροπρόθεσμα. Ε, υπάρχουν επίσης ε, ορισμένες ε, μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις περισσότερες από ό,τι έχουμε εμείς στη ΣΥΠΑ που θα μπορούσαν να ωφεληθούν από όλα αυτά. Η απουσία της εστίασης ε, στην βιομηχανική καινοτομία είναι αδύνατο σημείο σε πολλές στρατηγικές, εθνικές στρατηγικές ε, καινοτομιών. Τώρα, για το πώς οργανώνεται ένα project και τα, τα κονσόρτσια ε, στα πλαίσια του 2020, του Horizon 2020, μπορούμε να βελτιώσουμε τη διαφάνεια, ε, θα πρέπει να, ενδεχομένως να δημιουργηθεί ένα αρχείο, μια βάση δεδομένων, με ε, οτιδήποτε δημιουργήθηκε στα πλαίσια του FP7 και του Horizon 2020 και να μπορεί να υπάρχει πρόσβαση για να παίρνουν οι επιχειρήσεις την πληροφορία, αυξημένη ε, συμμετοχή επενδυτών στο, στη διαδικασία εμπορικής ε, εκμετάλλευσης γύρω από τα κονσόρσια. Μιλήσαμε επίσης και για την απλούστευση, απλοποίηση που είναι κλειδί θέμα, κύριο θέμα, ούτως ώστε να συμμετέχουν και αμερικανικές και άλλες εταιρείες ενεργά. Εμείς επίσης ε, ε, πριν από ε, ένα χρόνο μελετήσαμε στο Στάνφορ το FP7 και είχαμε και εταιρείε και καθηγητές από τη Δυτική Ακτή για να συμμετέχουν και μετά από μισή μέρα και με, με ένα πρόεδρο της, της συζήτησης για να ε, εξηγήσω και λιγάκι τα αμερικανικά δεδομένα και τις διαφάνειες. Οι περισσότεροι καθηγητές είπαν ότι είναι λίγα τα χρήματα και εξακολουθεί να θεωρείται πολύ δύσκολο να συμμετέχει κανείς στο FP7, στα και τα κονσόρτσια εκεί. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι θα έπρεπε να δημιουργήσουμε ε, ένα, ένα ρυθμό ε, δημιουργίας ανάπτυξης εταιρεία επιχειρήσεων ε, και αυτό που κάνουμε στα πανεπιστήμια, αυτό που γίνεται στα πανεπιστήμια είναι πολύ χρήσιμο για να ε, τεθούν ε, ρυθμοί ανάπτυξης επιχειρήσεων στο μηχανολογικό τομέα, στον τομέα διοίκησης επιχειρήσεων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και δημιουργεί στοιχεία που δεν χρησιμοποιούνται πολύ στην Ευρώπη. Ένα άλλο θέμα με αυτά τα κονσόρσια είναι ο κατακαιρματισμός της ε, πνευματικής ε, ιδιοκτησίας, ε, πράγμα που δημιουργεί επίσης προβλήματα. Είναι σημαντικό επίσης να συμμετέχει το επιχειρηματικό κεφάλαιο σε, όλα αυτά, σε όλες αυτές τις συζητήσεις και με το δίκτυο European Business Angels, το IBAN, ε, ενδεχομένως θα, μπορούσαν, ε, θα μπορούσε το δίκτυο Angels να αναλάβει ε, μεγαλύτερο ρόλο. το venture capital, η venture capital industry θα πρέπει να συμμετέχει και κάτι που δεν είναι στην ατζέντα καινοτομιών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί δεν αποτελεί ε, στοιχείο της εντολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επειδή είναι πολύ ευαίσθητο και δύσκολο θέμα. Νομίζω ότι η μεταρρύθμιση των πανεπιστημίων θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο της ατζέντα καινοτομία της Ευρώπης, των ευρωπαϊκών χωρών, γιατί αν δεν μπει κανεί μέσα στο πανεπιστήμιο για να αλλάξει την κουλτούρα του, αν δεν πιέσουν και οι φοιτητέ με τρόπο δραστήριο ε, μαζί με τους καθηγητές τους, αν δεν δημιουργηθούν ομάδες ε, μέσα στα ίδια τα ιδρύματα που θα πιέσουν για την πολιτισμική αυτή αλλαγή, δεν θα γίνει τίποτα. Χρειάζεται μια νέα κουλτούρα. Τα πανεπιστήμια θα πρέπει να κάνουν έρευνα με καινοτομία στις παρυφές. Δεν εξυπηρετεί πια. Ε, αυτό που βλέπω στο πρόγραμμα είναι ότι θα δημιουργήσει το Horizon 2021 σημείο καμπής. Ε, θα πρέπει να δώσει έμφαση ε, εγώ πιστεύω ότι αν δεν αντιμετωπίσουμε το θέμα της μεταρρύθμισης των πανεπιστημίων, δεν θα έχουμε την, ε, την αλλαγή αυτή που χρειάζεται. Ε, η Φιλανδία ε, αρχίζει να καταπιάνεται με αυτό το θέμα με άμεσο τρόπο. Το 2009 άρχισαν οι διαδικασίες, είναι νωρίς ακόμα, αλλά ε, κατάρτισαν οι Φιλανδοί μια στρατηγική για την μεταρρύθμιση των πανεπιστημίων. Ε, όλα τα δημόσια, τα κρατικά πανεπιστήμια μπορούν να δουλεύουν αυτόνομα και ανεξάρτητα και μπορούν έτσι να αλληλεπιδρούν πολύ καλύτερα και ευκολότερα με τις επιχειρήσεις, ε, να αποκομίζουν ε, δευτερεύοντα ωφέλη κλπ. Έφτασα στο τέλος της ομιλίας μου, περιμένω τις ερωτήσεις σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Grazie, dottor e, Iniziamo con eh, le domande. Voi avete tutti notato che abbiamo sforato i tempi. Πιέζει ο χρόνο, οπότε πρέπει να προχωρήσουμε ε, αμέσω στι ερωταπαντήσει. Ε, και βεβαίω ε, ο καθηγητής Λί ήρθε να μα μιλήσει από την Καλιφόρνια και εμείς έχουμε πάει, δεν έχουμε επισκεφθεί και μας έδωσε την ευκαιρία να ακούσουμε τι απόψει εκτός Ευρώπη. Και τώρα έχουμε δύο λεπτά για τον κάθε επόμενο αγορητή. Δύο ερωτήσεις έχω. Η πρώτη προς τον Υπουργό και το Υπουργικό Συμβούλιο με όλη την ευγένεια που επιτάσσει η περίσταση μετά από την παρέμβασή σας πρέπει να πω το εξή ότι είμαι απεσιόδοξο για το πώ θα διεξαχθούν οι διαπραγματεύσει μεταξύ Κοινοβουλίου και Υπουργικού Συμβουλίου. Θα ήθελα λοιπόν τι ερωτήσει να σα κάνω. Καταρχά, είναι κατανόητο το γεγονό ότι η Προεδρία τη Δανία ε, δεν έβαλε στην, επόμενο, στην επόμενη μερίσια διάταξη τους ε, κανόνες συμμετοχής. Γιατί βλέπουμε από μαθηματικής άποψης ότι έχουμε πολλούς αγνώστους. Δεν έχουμε ε, χρηματοοικονομικές προοπτικές. Ε, όλα αυτά έχουμε και ένα Υπουργικό Συμβούλιο που δεν έχει θέσει τα θέματα α, κανόνων συμμετοχής στο επόμενο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας. Μα τι θα αποφανθεί το Συμβούλιο. Θα παραμείνουμε όμοιροι των επόμενων δημοσιονομικών προοπτικής η δική σας Προεδρία και το γεγονός ότι αποφασίσατε να μην συζητηθούν αυτοί οι κανόνες αποτελεί απάρνηση των καθηκόντων σας και παρουσιάζει μεγάλες δυσκολίες σε ό,τι αφορά τις συνεργασίες μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Θα ήθελα λοιπόν να κάνετε κάποιες δηλώσεις από αυτού, ίσως και για το συνολικό θέμα, για το ότι Αν παραμείνουμε στα ίδια στοιχεία, μιλάμε για μια αύξηση 6 έως 7% το 2013. Και στην περίπτωση αυτή όμως δεν θα είμαστε σε θέση να πετύχουμε τους στόχους του 3% που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προς το ΑΕΠ. Δεν θα πετύχουμε λοιπόν τους στόχους αυτούς που έχουμε θέσει. Χρειάζεται λοιπόν μια νέα τοποθέτηση του Συμβουλίου. Μία ε, δεύτερη ερώτηση προς την Επίτροπο Κουίν. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερα στην εισήγηση που ακούσαμε, ακούσαμε θέματα της επιχειρηματικότητας σε ό,τι αφορά το, κεφάλαιο κινδύνου. Έχουμε και μία σχετικό, ένα σχετικό μέσο διευκόλυνσης ε, σε ό,τι αφορά τα δάνεια de facto πιο πολύ εστιάζεται στον ιδιωτικό τομέα και όχι τόσο στην επιχειρηματικότητα. Χρειάζεται λοιπόν μία επιπλέον διάσταση προκειμένου να λάβει τον πραγματικό ρόλο που της αρμόζει η επιχειρηματικότητα. Ποια είναι η δική σας θέση. Τελευταία ερώτηση για την διεθνή διάσταση, γιατί και αυτή αναφέρθηκε. το ερώτημα του κατά πόσον τα προγράμματα προϊόντων είναι αρκετά ελκυστικά. Έχουμε πάρα πολλούς στόχους που αναφέρθηκαν. Μιλάμε για αναδυόμενες οικονομίες, γειτονία, διεύρυνση, αναπτυσσόμενες χώρες. Κάνουμε αναφορά σε συγκεκριμένα πράγματα όπως κλινικές δοκιμές, βιοτεχνολογία και για προγράμματα για τους νεαρούς επιστήμονες το θέμα για την διεθνοποίηση είναι η στρατηγική διάσταση. Με ποιους εταίρους, υπό όρους θέλουμε συμμετοχή των εξαίρετων, των άριστων ε, περιφερειών και πώς θέλουμε όλα αυτά να τα, βελτιώ, να τα βελτιώσουμε. Ευχαριστώ. Κύριος Τσουκαλάς. Σε κυρία Πρόεδρε. Δύο ερωτήσεις ή μία ερώτηση στην κυρία Επίτροπο Τη συγχαίρω για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τη συνεργασία των διαρθρωτικών ταμείων με τα λοιπά ερευνητικά προγράμματα. Θα ευχόμουν αυτή η πρωτοβουλία της Επιτρόπου να πάρει συγκεκριμένη μορφή για τις χώρες εκείνες που καθυστερούν στην εφαρμογή της στρατηγικής της Λισαβόνας, όποια είναι και ο μηχανισμός στήριξης για την οικονομική στήριξη των ευρωπαϊκών κρατών. Κάτι τέτοιο μας χρειάζεται και για την έρευνα και για την τεχνολογία. Αν θέλουμε να υποστηρίξουμε την εξάπλωση της αριστείας σε όλη την Ευρώπη. Ευχαριστίες οφείλονται και στον κύριο Λί, εκπρόσωπο της Δημοκρατίας της Καλιφόρνια, ο οποίος μας είπε με την δική του προσωπική αντίληψη πώς βλέπει την Ευρώπη. Εάν κατάλαβα καλά, ο κύριος Λί μας είπε ότι η παντελής έλλειψη καινοτομικού πνεύματος μας φέρνει στη θέση του ανθρώπου του Νεάντερταλ που επειδή δεν μπόρεσε να καινοτομήσει καταφαγώθηκε από τον Κρόμανιόν. Τυχαίνει να είμαι της αυτής αντιλήψεως, ήθελα όμως να τον ρωτήσω πώς είναι δυνατόν σε μια χώρα, σε μια συμπολιτεία όπως είναι η Ευρώπη με διαφορετικό πολιτιστικό υπόβαθρο να αντιμετωπιστεί η έλλειψη της επιχειρηματικής καινοτομικότητας ή του venture capitalism το οποίο είναι ένα φαινόμενο που στην Αμερική άρχισε από το 1920 Πώς μπορούμε να διασκευάσουμε τα πανεπιστήμια μας όταν οι εταιρείε στην Αμερική και τα πανεπιστήμια βρίσκονται εδώ και δεκάδες χρόνια σε πολύ στενή επαφή. Πράγματι φαίνεται ότι αυτό πρέπει να γίνει, όμως θα περίμενα να μας πει αν βλέπει τον τρόπο να γίνει, γιατί από τις υποδείξεις του δεν καταλαβαίνω αυτό να γίνεται. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, λέει η Πρόεδρος και δίνω λόγο στον κύριο Κέλλη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τους ε, αγωγητές. Ήταν πάρα πολύ αξιόλογα τα όσα ακούσαμε και ε, νομίζω η Επίτροπος πολύ καλά μας τα είπε πρώτη-πρώτη. Ακριβώς. Θα πρέπει να δούμε πώς θα καλύψουν το χαμένο έδαφο σε σχέση με του ανταγωνιστέ μα, Κορέα, Ιαπωνία κλπ. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται σε σχέση με τη στρατηγική του 2020, συνέργεια και όλα αυτά. Επίση, ο Δόκτωρ Πέτερσεν μα είπε για τα προϊόντα και την αγορά, τα νέα προϊόντα που πρέπει να μπαίνουν στην αγορά και επίση ο καθηγητής Λίμα τα είπε καλά. Τον ευχαριστώ για τα καλά λόγια για την χώρα μου και ήμουν τυχερό. Είχα την τύχη να βρίσκομαι πέρσι. Εγώ με τον Πίτερ Σκίνερ στην Silicon Valley. Το θέμα είναι πώς θα μεταλαμβαδεύσουμε την εκεί επιτυχία στην Ευρώπη. Για πετε μου, κυρίω η Επίτροπο, τι λέτε για αυτά που είπε ο Δόκτωρ Λί. Όσον αφορά τις απασχόληση. νέα προϊόντα, αυτά είναι τα κριτήρια τη επιτυχία μα και όχι το πόσα χρήματα δίνουμε στην έρευνα. Πώς επομένως θα μπορέσουν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να δημιουργήσουν την κρίσιμη μάζα ερευνητών. Τι να κάνουμε και στο 2020 να μπορούμε να πούμε ναι. Πετύχαμε τους στόχους μας για έρευνα ανάπτυξη. Τους στόχους μας για νέα προϊόντα. Και όσον αφορά την απασχόληση πιάσαμε τους στόχους μας. Να μπορούμε αυτά όλα να τα πούμε το 2020. Ευχαριστώ. Γκλάντα. Σας ευχαριστώ. Επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Dr. Burton Lee για τις μεγάλες αλήθειες που είπε και πολλά από αυτά θα πρέπει να τα σκεφτούμε. Δύο ερωτήσεις έχω να κάνω προς την Δανική Προεδρία και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα να συμφωνήσω με τον συνάδελφο Έλα το συγκεκριμένο ερώτημα που έχω να θέσω είναι το εξή. Όταν λέτε ότι ο προπολογισμό θα αποφασιστεί από την Ιρλανδική Προεδρία, το θέμα είναι κατά πόσον μιλάμε και για το πρόγραμμα Ορίζοντες 2020 ε, γιατί αν είμαστε ειλικρινείς φυσικά μπορούμε κάθε μέρα να ζητάμε αύξηση του προπολογισμού για τα προγράμματα αλλά Νομίζω ότι δεν θα περάσουν αυτά στο Συμβούλιο. Θα πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή να αποφασίσουμε πού θα κάνουμε περικοπές, ακόμα και μέσα στο ίδιο το πρόγραμμα. Και θα ήθελα να ακούσω προτάσεις από το α, Συμβούλιο και όχι μόνο εμείς, το Κοινοβούλιο, να γίνουμε οι κακοί που θα προτείνουμε περικοπές, να δούμε το α, Τεχνολογικό Ινστιτούτο προκειμένου να αποφεληθεί στο κοινοβουλιο να γινουμε οι κακοι που θα προτεινουμε περικοπες να δουμε το τεχνολογικο ινστιτουτο προκειμενου να αποφεληθει το προγραμμα Μαρικιουρή, για παράδειγμα, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλουμε να δημιουργήσουμε αυτή τη σκάλα προς την αριστεία και γίνονται απόπειρε να συνδυαστεί η περιφερειακή πολιτική με την πολιτική για την ε, έρευνα. Υπάρχει συντονισμός όμως των μέσων αυτών. Μπορούμε δηλαδή να εφαρμόσουμε ε, υποχρεωτικά μέσα διαφορετικά σε συνδυασμό με τα μέσα για την ε, έρευνα, γιατί μου λείπει αυτή η εγγύηση από αυτά που μας ανέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Τσουμπίχ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι η συζήτηση για τα μέσα αποτελεί ένα βασικό θέμα, γιατί ιδιαίτερα στο σημερινό σύστημα αντιμετώπισης του χρέους ε, στην Ευρώπη δεν είναι τα πράγματα ρόδινα για τα προγράμματα αυτά. Κυρία Επίτροπε, ίσως ο συνάδελφός σας για τη φορολογία θα μπορούσε στο Small Business Act να δώσει τη δυνατότητα να υπάρξει ένα πρόγραμμα φορολόγησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με το βέλτιστο δυνατό τρόπο. Αφενός, για παράδειγμα, στα, στα λογιστικά συστήματα να υπάρχουν κάποιες επιδοτήσεις για την έρευνα, να δοθούν κίνητρα προκειμένου οι επιχειρήσεις να μπορούν να διαμορφώσουν ε, ίδιο κεφάλαιο, κεφάλαιο κινδύνου για να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους, αλλά όλα αυτά να μπορούν να τα έχουν συγκεντρώσει προτού τα αφιερώσουν σε τέτοιους σκοπούς. Ίσως να υπάρχει και ένας ε, ενιαίος φόρος σε κάποιες περιπτώσεις. Ε. Όλοι όσοι δραστηριοποιούνται στο τομέα της έρευνας να μην πληρώνουν φόρο εισοδήματο. Να υπάρχουν τέτοιες ελαφρύνσεις προς τις επιχειρήσεις προκειμένου να μπορούν παράλληλα να δίνουν υψηλούς μισθούς. Υπάρχει καν αυτή η έννοια της αποτελεσματικότητας της φορολογίας. Ή μήπω θα μπορούσαμε τον οδικό χάρτη για το 2020 να τον διαμορφώσουμε προ την κατεύθυνση τη βέλτιστη αυτή φορολόγηση. Ευχαριστώ. Η κυρία Μαρκή. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, κύριοι και κυρίε του πάνελ, ευχαριστούμε για όλα όσα μα είπατε. Θα ήθελα να απευθυνθώ στον καθηγητή Μπέρτον Λί, τον οποίο έχουμε ξανασυναντηθεί στην Silicon Valley. Και με εντυπωσίασε αυτό το οποίο είπε για την καινοτομία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε ανοιχτοί. Δηλαδή, να έχουμε κάποιους που όντας πάνω από 80 και αυτοί να συμμετέχουν. Δηλαδή να μην απευθυνόμαστε μόνο στους νέους. Όλους, όλους να θέλουμε να καλύψουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, να καλυφθούν όλες οι ηλικιακές κατηγορίες. Επίσης, παρακαλούμε, πέστε μας. Τι μπορούμε να κάνουμε για την πολιτική της Ένωσης. Ας πούμε, έχουμε τομιακή προσέγγιση στις 100 θεματική. Ε, όμως ε, η Ευρώπη κυρίως ε, ε, ε, υιοθετεί την οπτική γωνία των αλλαγών της κοινωνίας, της προκλήσεων της κοινωνίας, societal challenges. Κύριε Λί, επίσης μας είπατε για τους στόχους. Έχετε κάποιο παράδειγμα ο, κατά, από τη δική σας χώρα που πετύχατε κάποιους στόχους. για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων. Περισσότερο κρατάω το ενδιαφέρον σας στο λογισμικό και είπατε ότι δεν προσέχουμε όσο πρέπει το, το λογισμικό. Όμως χρειαζόμαστε την προσοχή μας να τη και αλλού. Δεν μπορούμε να είμαστε όλοι οι ειδικοί υπολογιστέ. Τι γίνεται, δεν μπορούμε να, συνδυάσουμε περισσότερο για να έχουμε έτσι ένα μείγμα πολιτική, περισσότερο, περισσότερου στόχου. Ευχαριστούμε. Κυρία Γκουτιέρα, σα ευχαριστώ πολύ. Κάτι το οποίο σήμερα με απασχολεί είναι το εξή. Ο κύριος Λί μίλησε για έννοιε και όχι για συγκεκριμένα πράγματα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να προβληματιστούμε όσον αφορά την έννοια της Ευρώπης της καινοτομία, γιατί πρόκειται για αυτή την κουλτούρα της καινοτομία, της ε, αξιολόγηση και αξιοποίηση. Με τέτοιο τοπίο θα βοηθήσουμε την ανανέωση και την έρευνα. Μιλούμε για τομιακές πολιτικές και εδώ συνήθως κάνουμε τροπολογίες σκόρπιες. Αυτό το οποίο θέλουμε είναι το τι θα κάνουμε για να βοηθήσουμε και τις μητριότητες. Άρα πρέπει να αλλάξουμε μοντέλο συνήθειες. Με αυτό το πνεύμα θα ήθελα να πω ότι αν δεν αλλάξει το πανεπιστημιακό μας πρότυπο να έχουμε σύστημα αξιολόγησης και όχι λογοδοσία. Έχουμε ολοκληρωμένη προσέγγιση και όχι κατάτμιση προσεγγίσεων. Για την κύριε Επιτρόπο και μετά για τον κύριο Ελία. Εάν επομένω δεν κάνουμε μια εκβάθρα αναλλαγή, πώς θα είναι δυνατόν κύριε Επίτροπε να τολμήσουμε και έχετε τη βοήθεια του Κοινοβουλίου να προβούμε σε κάποιον έλεγχο των προβλημάτων που έχουμε στα κράτη, στα πανεπιστήμια και να προταθούν λύσεις. Να υπάρχει τόλμη να γίνουν αυτές οι αλλαγές. Να κάτσουμε να αξιολογήσουμε τι ισχύει, τι γίνεται με τα πανεπιστήμια και να επικρατήσει επιτέλους αξιοκρατία. Έτσι να ανοίξουν οι πύλες των πανεπιστημίων. Κύριε Λία, για σας. Πώς θα αλλάξουμε επομένω την κουλτούρα, πώς θα αλλάξουμε το πρότυπο για να πάμε σε μεταρρυθμίσεις. Ας πούμε το λέιζερ. Είναι πολύτιμο. Είδατε πώς γίνονται οι χειρουργικέ συμβάσει με το λέιζερ. Μπαίνει το λέιζερ ει βάθος και κάνει την εγχείρηση. Τόια. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστούμε όλους όσους έλαβαν το λόγο. Έχω μια πρώτη ερώτηση προς την Επίτροπο. Ακούσαμε το πόσο σημαντικό είναι το να έχουμε εκμετάλλευση εμπορική των αποτελεσμάτων της έρευνας και για πέστε μας τι θα μπορούσε να γίνει ούτως ώστε αυτή η αρχή να ισχύσει και στην Ευρώπη. Νομίζω ότι υπάρχουν μελέτες που είναι σημαντικές και επομένως αξίζει να βοηθηθεί η πρόθεση των προϊόντων που βγαίνουν στην Ευρώπη κατόπιν έρευνας ευρωπαϊκής. Δεύτερον, συνέργεια, συντονισμός, συμπληρωματικότητα. Τι λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τους πόρους της, ε, του Ταμείου Συνοχής και από την άλλη μεριά τους πόρους για το Horizon 2000. Πώς θα μπορούσαμε να έχουμε υποδομή που να βοηθά την έρευνα. Θα μπορούσαμε να έχουμε συμπληρωματικά προγράμματα, διατομιακά και να εκμεταλλευτούμε επομένως αυτούς τους πόρους. Θα πρέπει να συμφωνεί το κοινοβουλίο όταν λάβουμε τι ε, προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα πρέπει να προχωρήσουμε προ μια διαδικασία συναπόφαση για τη σχετική έγκριση αυτών των προτάσεων. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τους ομιλητές για τις πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις τους σε ό,τι αφορά το μελλοντικό μας έργο, αλλά θα ήθελα να δράξω αυτή την ευκαιρία για να συνεχίσω αυτή τη σύγκριση μεταξύ ΙΠΑ και Ευρώπης. Θα ήθελα δύο ερωτήσεις να κάνω ως προς αυτό. Ο κύριος καθηγητής Λί ανέφερε στο τέλος ότι δεν είναι δική μα ευθύνη να φροντίσουμε τις μεταρρυθμίσει των πανεπιστημίων. Παρ' όλα αυτά όμως αυτό επηρεάζει τη διαμόρφωση του προγράμματο μα σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα Horizon. Γιατί μέσω των προγραμμάτων αυτών μπορούμε να φροντίσουμε να υπάρχει πιο ανοιχτός χαρακτήρα στα πανεπιστήμια. Έχετε συγκεκριμένες προτάσεις λοιπόν πώς μπορούμε στο μελλοντικό μας έργο ως εισηγητές να συμβάλλουμε προκειμένου το πρόγραμμα Horizon 2020 να διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο προκειμένου να δοθεί στα πανεπιστήμια και στις τεχνικές σχολές ανοιχτός χαρακτήρας. Αυτό ήταν η πρώτη ερώτηση. Η δεύτερη ερώτηση. Ακούσαμε τα περί Silicon Valley. Αναφερθήκατε στη Σουηδία, στη Φιλανδία και σε άλλες χώρες. Το επόμενο ερώτημα λοιπόν είναι το εξής. Αν στην Ευρώπη μπορούμε να δώσουμε και να ενισχύσουμε την ε, συνολική καινοτομία και την έρευνα, αν αφενός προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε με μονομένα συστήματα σε διάφορες περιφέρειες. Για παράδειγμα, αναφερθήκατε σε κάποιες περιοχές που είναι ήδη πολύ δυναμικές σήμερα. Αλλά αυτό είναι το πιο σωστό ή μήπως θα έπρεπε μέσω του προγράμματος ε, Horizon 2020 να υπάρχει ανταλλαγή, συνεργία μεταξύ των διάφορων τομέων στην Ευρώπη. Πώς θα είμαστε πιο αποτελεσματικοί θεωρείτε για να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, τι θα μας προτείνατε, τι θα μας συστήνατε, ποιος θα ήταν ο καλύτερος συνδυασμός, θεωρείτε. Ευχαριστώ. Και τώρα... Θα πρέπει, δυστυχώς, να παρακαλέσω και την κυρία Επίτροπο να τηρήσει το χρονικό όριο και τους εκπροσώπους του Συμβουλίου και του καθηγητή Λί. Έχετε το λόγο. Θα ήθελα λοιπόν να είμαι όσο πιο σύντομη γίνεται για το ερώτημα του κύριου Έλλη και πολύ λυπάμαι που δεν είναι εδώ. Α, είστε εδώ, μάλιστα. Πολύ ωραία. Αλλάξατε, αλλάξατε θέση. Είχα σημειώσει το έδρανό σα για το θέμα του κεφαλαίου κινδύου. Όπως ξέρετε, το μέσο για την διευκόλυνση ε, είναι πάρα πολύ κατέληξε στα ίδια συμπεράσματα ότι τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ε, ε, έχουν τεράστια μόχλευση και έχουν βοηθήσει πάρα πολύ τις επιχειρήσεις. Το Δεκέμβριο, νομίζω, με τον Φίλιπ Μάιστατ υπέγραψα μία συμφωνία για τροποποίηση της ε, Συμφωνίας Συνεργασίας με τρεις σκοπούς. Να δώσει στο RSSF μεγαλύτερη μόχλευση, σε ό,τι αφορά την κατανομή των πόρων που διατίθεται, που είναι πολύ σημαντικό. Κατά δεύτερον, να επιτρέψει στη Συμφωνία Συνεργασίας να αναφερθεί σε θέματα υποδομών ερευνάς και προκειμένου το Ταμείο Επενδύσεων να διαθέσει δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γιατί αυτές είναι που είναι κρίσιμες σε αυτή τη φάση του RSFF. Γιατί επικεντρωνόμαστε ως τώρα σε πολύ μεγάλα έργα και μεγάλες εταιρείες. Αυτά είναι τα προγράμματα. Ξέρετε τι θα γίνει και μετά μέσα για το χρέος. Για την εσωτερική διάσταση τώρα, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσουμε τα συμφέροντα για τον κύριο Τσουκαλά και τον κύριο Γκλάντε. Μιλήσατε για τη διάδοση της αριστείας και την ε, διεύρυνση της συμμετοχής. Ξέρω ότι ο Γενικός Διευθυντής Σμιτς μίλησε για το θέμα αυτό το πρωί. Δεν πρόκειται λοιπόν να επαναλάβω τα όσα είπε. Έχετε και δύο δίκιο όμως ότι η συνέργεια μεταξύ των διαφορετικών ταμείων και του προγράμματος Horizon 2020 θα είναι κρίσιμη για την ε, διάδοση της αριστείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θεωρώ ότι τα διευθυντικά ταμεία εμπλέκονται στην ανάπτυξη των υποδομών, στην, ε, στο hardware αν θέλετε και το Horizon 2020 θα ανταποκριθεί αναγνωρίζοντας την αριστεία των υποδομών αυτών και κατά δεύτερον χορηγώντας ε, τους πόρους που χρειάζονται για παράδειγμα για να χρησιμοποιήσουν οι καθηγητές τις υποδομές αυτές και να δημιουργήσουν την αριστεία που επιθυμούμε. Κύριε Γκλάντε, α, συγγνώμη, ο κύριο Κέλλη και η κυρία Κουτιέρε Κορτίνε μιλήσανε για τα πανεπιστήμια και τον εξυγχρονισμό του. Φυσικά και οι δύο σημειώσατε ότι αυτό δεν είναι στις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ξέρετε όμως ότι η Επίτροπος Βασιλείου έχει, υπογρα... έχει ε, δημοσιεύσει μια ανακοίνωση για τα πανεπιστήμια και το έχουμε πει σε πολλαπλές περιπτώσεις ότι θα πρέπει κατεπηγόντως να εξυγχρονιστεί το πανεπιστημιακό σύστημα, γιατί θεωρώ ότι έχει παραπάει πια αυτή η ακαδημαϊκή φούσκα. Έχει διτηρηθεί υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα. Χρειάζεται συνεργασία με τη βιομηχανία. Έχουν περάσει αυτές οι ημέρες. Αν θέλουν τα πανεπιστήμια να διακρίνονται, θα πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία τη βιομηχανική. Κοιτώντας ένα σύστημα το οποίο κοιτάμε εμείς στο ευρωπαϊκό χώρο ερευνών, θα πρέπει να είναι σαφές ότι η πρόσληψη στα πανεπιστήμια θα πρέπει να γίνεται με διαφάνεια και με αξιοκρατικά κριτήρια. Όλοι ξέρουμε ότι αυτό δεν συμβαίνει σε σημαντικό αριθμό των πανεπιστημίων σήμερα. Αυτή είναι λοιπόν η πρόκληση για τα κράτη-μέλη και πρόκειται για μια πρόκληση την οποία σκοπεύουμε να θέσουμε προς τα κράτη-μέλη και υπολογίζουμε στη βοήθειά σας. Γιατί πρόκειται για το ένα θέμα το οποίο μου ανέφεραν οι νεαροί ερευνητέ στο Ιβοστόνι. 95% εξ αυτών ήταν Ευρωπαίοι που είχαν φύγει από την Ευρώπη, αλλά όλοι ήθελαν να γυρίσουν στην Ευρώπη. Αλλά μου διευκρίνησαν ότι για να γυρίσουν στην Ευρώπη χρειάζονταν ένα διαφανές αξιοκρατικό σύστημα πρόσληψης στα πανεπιστήμια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κύριε Ρούμπιχ, για το φορολογικό σύστημα θα ξέρετε καλά ότι οι φορολογικέ αλλαγέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μάλλον δύσκολες και συμβαίνουν μόνο με ομοφωνία 27 κρατών μελών. Κάποιοι μπορεί να επιθυμούσαν κάτι διαφορετικό, έτσι έχει η κατάσταση όμως σήμερα. Νομίζω όμως υπάρχουν πολύ καλά παραδείγματα σε κάποια κρατημέλη όπου έχει αλλάξει το φορολογικό σύστημα προς όφελος της επένδυσης στην έρευνα και την κοινοτομία. Νομίζω ότι τα κράτη-μέλη που δεν το έχουν πράξει αυτό ακόμη θα μπορούσαν να εξετάσουν τις προτάσεις αυτές και φυσικά στο κράτος μέλος που γνωρίζω καλύτερα από όλα εισήχθη πρόσφατα αυτή η νομοθεσία. Νομίζω ότι ήταν πολύ θετικό αυτό για την κυρία Τόγια τώρα. Καταρχάς σε ό,τι αφορά το Europe Exploitation προτάθηκε από την ομάδα υψηλού επίπεδου, για τις τεχνολογίες υψηλού επίπεδου. Δεν το δεχτήκαμε γιατί δεν πιστεύουμε καταρχάς ότι θα πρέπει να υπάρχει η εκμετάλλευση αυτή πρώτα στην Ευρώπη ως κανόνα. Αν υπάρχει κάποιο στρατηγικό συμφέρον, αν υπάρχει μια μεγάλη ευρωπαϊκή επένδυση, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε το ζήτημα της πρώτης εκμετάλλευσης στην Ευρώπη κατά περίπτωση, αλλά πάντα περηφανευόμαστε ότι η έρευνα και η καινοτομία είναι στην Ευρώπη η πιο ανοιχτή στον κόσμο και αυτό θα θέλαμε να συνεχιστεί. Και στο σημείο αυτό θα κλείσει ο Πρόεδρος Ατόρη. Ευχαριστούμε πολύ. Μπορείτε να απαντήσετε σε όλα. Και τώρα ο Δόκτωρα Πέτρας έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να είμαι και εγώ όσο γίνεται πιο σύντομος τον κύριο Γκλάντα ε, και όποιον άλλο με ρώτησε γιατί θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για την υπόθεση του Horizon 2000, 2020. Φυσικά και η συμμετοχή είναι κάτι πάρα πολύ βασικό και οι σχετικοί κανόνες οπότε όλα αυτά πρόκειται να συζητηθούν και στο επόμενο Συμβούλιο. Τώρα, ε, βρισκόμαστε στη φάση κατά την οποία όλα τα κράτη-μέλη ε, θα πρέπει σελίδα-σελίδα να αναλύσουν ε, το πακέτο, τη δέσμη των μέτρων και έτσι να μπορέσουμε, ελπίζω, μέχρι το επόμενο Συμβούλιο, δηλαδή τέλη μαΐου να καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία σε σχέση με το επόμενο πρόγραμμα πλαίσιο θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ λογικό να συζητηθεί η αρχιτεκτονική του προγράμματο και τα θέματα σχετικά με του πόρου θα συζητούν αργότερα. Συμπερασματικά πρέπει να σα πω επίση ότι μα ενδιαφέρει πάρα πολύ το να έχουμε αγαστή συνεννόηση και διάλογο με το Κοινοβούλιο. Ήδη έχουν γίνει κάποιε διαβουλεύσει. Στην Κοπενχάγη επίση πήγε πάρα πολύ καλά το άτυπο συμβούλιο και όπως είπα στην εισαγωγή, την αρχική μου εισήγηση, ελπίζουμε ότι θα, προ, θα, θα, το έδαφος, θα εξελίσσουμε τις ε, διαφωνίες και θα τα πάμε καλά ενώ της συνάντησης των αρχών Μαΐου και τη συμφωνία του να πετύχουμε μέχρι το τέλος του Μαΐου οπότε δικαιολογημένα νομίζω είμαστε αισιόδοξοι και φιλόδοξοι Ευχαριστούμε καθηγητά Ευχαριστώ Συγγνώμη αν ε, παραλείψω να απαντήσω σε κάποιον. Πιστεύω, κύριε Έλερ, ε, ρωτήσατε για το εύρος στο οποίο διδάγματα ε, από την αμερικανική εμπειρία μπορούν να υλοποιηθούν. Ήδη κάποια σημαντικά στοιχεία ε, και από τη ΣΥΠΑ και από τον Καναδά έχουν ληφθεί υπόψη. Ε, πολλή σκέψη και οργάνωση έχει δοθεί σε αυτή την προσπάθεια, οπότε ήδη συμβαίνουν όλα αυτά ε, στα πλαίσια της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας, δηλαδή παίρνουν τα διδάγματα. Η αφορά τώρα την ε, προσέγγιση. Ε, δεν, ε, ελπίζω να μην έδωσα ένα αρνητικό μήνυμα σε σχέση με αυτά που γίνονται. Είναι πολύ σημαντικό να αλλάξει η κουλτούρα στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια μπορούν αντιπροσωπείες φοιτητών, ε, καθηγητών, 20-30 ε, κάθε φορά δύο φορές το χρόνο, μπορούν να έρθουν για μία εβδομάδα τουλάχιστον ε, στην Silicon Valley να επισκεφθούν τα πανεπιστήμια Stanford, Berkeley, να δουν τι γίνεται στο Stanford, να πάνε μέσα στο πανεπιστήμιο να δουν πώς λειτουργεί, στο Berkeley επίσης, γιατί αυτό επηρεάζει πάρα πολύ. Επίσης, ε, τα ανοιχτά, ε, πολύ ανοιχτά πανεπιστήμια που είναι τα φιλανδικά και κάποια βρετανικά προσκαλούν επιχειρήσεις ε, ή στα πανεπιστήμια ή σε κάποιες σχολές συγκεκριμένα ανάλογα με τον τομέα και αυτό επίσης είναι πολύ θετικό. Τώρα στον κύριο Κέλλη για τα νέα προϊόντα και θέσεις εργασίας η πολιτική καινοτομιών έχει κάποια έλλειψη σε ένα προγραμματικό επίπεδο. Τα προγράμματα είναι της Κομισιόν ή διεθνικά προγράμματα. Υπάρχουν προγράμματα που λείπουν όμως, όπως για τη σχεδιασμό προϊόντων. Δεν είναι στην ατζέντα των πανεπιστημίων επίσης. Ε, πολλές φορές ε, ε, λειτουργούν σε χαμηλότερο επίπεδο. Δηλαδή πολλά πανεπιστήμια δεν περιλαμβάνουν ε, σχεδιασμό προϊόντων. Αυτό σημαίνει διαφορετική κουλτούρα διαφορετική συνειδητοποίηση του πώς γίνεται στο MIT, στο Stanford ε, ο σχεδιασμός των προϊόντων. Στον κύριο Μέρκης, στην κυρία Μέρκης. Ε, εγώ στα 48 και στα 50 ε, ολοκλήρωσα ε, επιμέρους ε, ε, σπουδές και εξειδίκευση. Αυτό το παίρνουμε πολύ σοβαρά. Δεν μπορούσα να το κάνω στην Ευρώπη φαντάζομαι. Γυναίκες επιστρέφουν στις σπουδές αφού κάνουν τα παιδιά τους στην ηλικία των 40 ετών πολλές φορές. Έτσι υπάρχει μόχλευση του δυναμικού του καθενός σε προσωπικό επίπεδο. Ε, επίσης παραδείγματα από τις είπα για ε, νέες επιχειρήσεις ή προγράμματα. Κάποια πανεπιστήμια στις μεσοδυτικές πολιτείες το κάνουν αυτό. Δεν είναι πολύ διαδεδομένο. Στην Εμπράσκα, ε, πολιτείες που έχουν περισσότερες δυσκολίες στον τομέα αυτό, αρχίζουν όμως νέες επιχειρήσεις. Τώρα για το λογισμικό, στους τομείς ICT, και σε άλλους τομείς, στην υγεία για παράδειγμα, το λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε κάθε τομέα της ζωής και σε κάθε προσπάθεια. Ε, στο ε, ε, Γκουτιέρες Κορτίνες είναι καλό αυτό που είπατε για την αξιολόγηση πολλές φορές λέτε υπάρχει μια κουλτούρα στην Ευρώπη. Εμείς μιλάμε για σχεδιασμό και ε, δημιουργία κουλτούρας στις επιχειρήσεις, στις περιοχές. Γιατί να μην μιλήσουμε για αυτά που προϋποτίθενται για να αλλάξει η κουλτούρα ώστε να δημιουργηθούν πιο καινοτόμα ιδρύματα και επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Το Google, με αποφάσισε τι κουλτούρα θέλει ε, τι ανθρώπους χρειάζεται γι' αυτό, τι κίνητρα, τι συστήματα ε, υποβολής εκθέσεων και αναφορών, ε, ούτως ώστε να έχει την καλύτερη καινοτόμο κουλτούρα. Και στην Silicon Valley ισχύει αυτό. Και γι' αυτό το Google μπήκε σε καινούργιες αγορές με συνεχείς και αδιάλειπτους ρυθμούς. Μπορεί έτσι να αλλάξει η κουλτούρα τους. Για τον κύριο Τζόνσον δεν γνωρίζω το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλευτικό Σύστημα τι μπορεί και τι δεν μπορείτε να κάνετε, αλλά κάποιος πρέπει να βγει μπροστά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και να χτυπήσει συναγερμό υπέρ της μεταρρυθμίσης των πανεπιστημίων. Μπορεί κάτι να το κάνει... Μπορεί, ε, τα κοινοβούλια θα πρέπει να το κάνουν αυτό το πράγμα ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να παίξουν ηγετικό ρόλο ούτως ώστε να αναβαθμιστεί αυτό το θέμα και να αναδειχθεί σε πολιτικό επίπεδο. Επίσης, πώς θα βελτιώσουμε την ποιότητα της έρευνας στα ε, ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Κάτι που παρατήρησα σε κάποια μικρότερα πανεπιστήμια ε, είναι ότι πρέπει να μπει κανεί στις επιχειρηματικές διαδικασίες. Τα πανεπιστήμια να μπουν στις διαδικασίες, τα πολωνικά πανεπιστήμια, για παράδειγμα δεν ξέρουν τι γίνεται εκτός Πολωνίας όταν είναι μικρά τα πανεπιστήμια. Ε, περιορίζονται στη γνώση των καθηγητών από τον περιορισμένο κύκλο τους. Δεν έχουν ευρύτερο σημείο αναφοράς. Πρέπει λοιπόν να προσεχθεί πολύ το ζήτημα της επιλογής των ερευνητικών θεμάτων, η ερευνητική στρατηγική, μέσα στα πανεπιστήμια, από τον Πρίτανη μέχρι τον, τους καθηγητές και πώς θα επιλεγούν καλά θέματα για την έρευνα. Επίσης, ε, σε επίπεδο ε, εθνικών ερευνητικών ιδρυμάτων θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία ε, με επιστημονικά ιδρύματα, γιατί υπάρχει πολλή δυνατότητα ανταλλαγής συμβουλών για αυτό που είναι σημαντικό στην έρευνα κάθε φορά. Έτσι λειτουργούμε στη ΣΥΠΑ. Ε, το θέμα των αρμοδιοτήτων ε, θα πρέπει να το δούμε και στην, ε, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε <clears throat> τι αρμοδιότητες έχουν τα πανεπιστήμια, ο πρίτανης, τι εκπαιδευτικές ανάγκες υπάρχουν αυτό πρέπει να βελτιωθεί η διαχείριση γύρω από την έρευνα, την καινοτομία, γιατί τα περισσότερα πανεπιστήμια δεν γνωρίζουν τι γίνεται στις Ηνωμένε Πολιτείε ή σε άλλες περιοχές του κόσμου. Αυτό πρέπει να, να... να αλλάξει. Ευχαριστούμε, λέει Πρόεδρος. Ε, ευχαριστούμε όλους τους ε, αγορητές, ευχαριστούμε το Συμβούλιο, ευχαριστούμε την κυρία Επίτροπο, ευχαριστούμε τον καθηγητή Λί έχουμε διαθέσει πάρα πολύ σε σχέση με, τα, με, το πρόγραμμά μας και σας ευχαριστούμε χαιρετώντας σας. Ευχαριστώ. Πρέπει να αρχίσουμε τη συνέχεια των εργασιών μας. Παρακαλώ. Και αρχίζουμε δίνοντας το λόγο διακόπτη πρόεδρος συνεχίζει δίνοντας τον ε, λόγο για να κάνετε σχετική εισαγωγή στην ε, Μαρία Νταγράφια Καρβάλιο. Ευχαριστώ πρόεδρε, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Αρχίζω αναφέροντάς σας ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη μου χαρά να κάνω την εισαγωγή σε αυτό το πάνελ για ένα σημαντικό ε, ε, θέμα όπως είναι η ΜΜΕ σε σχέση με την βιομηχανία. Κάτι για τη σημερινή συγκύρια πολύ σημαντικό. Η συμμετοχή στα αρνητικά προγράμματα μας έχει δείξει την τάση ε, αυτήν τα τελευταία χρόνια ούτω ώστε να υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα αποτελέσματα της έρευνας που χρησιμοποιούνται ε, στην ε, διαδικασία αυτή σε σχετιστήτες χώρες και οπότε τα προγράμματα αυτής της κατασκευαστικής διαδικασίας ε, θα πρέπει να εξεταστεί τι γίνεται όταν πηγαίνουν στην Ευρώπη για κατανάλωση. Έχουμε μόνο μια σειρά στόχων που θα πρέπει να πετύχουμε. Την συμμετοχή των καινοτόμων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ε, να αναβαθμιστεί σε σχέση με το Horizon 2000. Θα πρέπει επίσης να τονωθούν οι ιδιωτικές επενδύσεις και επίσης ε, να δούμε τι θα γίνει και με την αγορά, διότι σε σχέση με αυτούς τους στόχους έχουμε κάποιες προκλήσεις που θα πρέπει να προσέξουμε επιγόντως και θα σας πω ποιες είναι αυτές πρώτα-πρώτα πώς θα εξασφαλίσουμε το πώς βλέπουμε εμείς τον ρόλο μας ως πρωτοπόροι ε, και πώς θα μπορούμε να δούμε αρκετά ε, ε, ευρέως τα πράγματα και για την βιομηχανία αλλά και για τους άλλους πυλώνες. Για το ορίζον 2020 θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την πρωτοπορία μας στον τομέα της βιομηχανίας και επίσης θα πρέπει να βλέπουμε υπόψη τις προκλήσεις αλλά και την αριστεία. Κάτι άλλο το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει είναι πώς το Horizon 2000 θα καλύψει όλη τη διαδρομή από έρευνα μέχρι αγορά. Ε, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ όρημη η αντιμετώπιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά δεν μας λέει αρκετά πάνω σε αυτό όσον αφορά το τελευταίο κομμάτι της αλυσίδας της καινοτομία και θεωρούμε ότι θα πρέπει να δοθεί ξεκάθαρος σαφής ο ορισμός τι γίνεται με τα πιλωτικά προγράμματα, τα προγράμματα ναυαρχίδες κλπ. Και να δούμε πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε βήματα προόδου προς την εμπρός. Επίσης έχουμε διάφορα μέσα πολιτικής. Κατά τη γνώμη μου έχουμε υπερβολικά πολλά και θα πρέπει να απλουστεύσουμε τα μέσα που έχουμε διαθέσή μας και κατόπιν να, να διαλέξουμε εκείνα τα οποία θεωρούμε ότι είναι τα πιο δόκιμα για την επίτευξη του στόχου. Να σας πω και κάποια παραδείγματα, έχω τα GTIs, GPIs, PPP και όλα αυτά κλπ. Οπότε θα πρέπει να δούμε τι είναι το πιο χρήσιμο, το πιο δόκιμο για τον στόχο μας. Επίσης, τι γίνεται με την ε, ε, χρηματοδότηση, γιατί απαιτούνται πολλά λεφτά. Και επομένως χρειάζεται μια πολυκλαδική προσέγγιση και να δούμε ποια διευθυντικά ταμεία έχουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο για να εξασφαλίσουμε συμβατότητα με το πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων που ισχύει. Περιμένω πώς και πώς να ακούσω τις ιδέες σας. Πώς θα ανταποκριθούμε σε αυτές τις προκλήσεις. Άλλωστε έχω αναλάβει και μια έκθεση για την ε, υλοποίηση του προγράμματος Horizon 2020. Με ενδιαφέρει επομένω ακόμη περισσότερο το τι θα μας πείτε, πώς θα απαντήσετε σε αυτές τις ερωτήσεις. Και έτσι θα με βοηθήσετε πάρα πολύ σημαντικά στην έκθεση που έχω, άλλωστε ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες θα σε ευχαριστούμε και περιμένω να συνεχιστεί η σημαντική μας ε, εκδήλωση απόψινή. Πείτε σκηνό, έχετε το λόγο, λέει Πρόεδρος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να είμαι το πιο δυνατόν σύντομο. Νομίζω ότι η Ευρώπη καμιά φορά κινείται σε κύκλου, μιλώντα για βιομηχανική ε, χρηματοδότηση για τι μικρέ επιχειρήσει και η ηγεσία ουσιαστικά προέρχεται από άλλο τμήμα του κόσμου ενώ θα έπρεπε ουσιαστικά να την αναπτύσσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε τα καλύτερα χρηματοοικονομικά μέσα και ειλικρινά έχουμε παράλληλα και τα χειρότερα χρηματοοικονομικά μέσα και το είδαμε αυτό στην κρίση. Αυτό το μείγμα ε, μας έκανε όλους να καταδικάζουμε τις οικονομικές υπηρεσίες. Υπάρχει λοιπόν αυτή η δυσκολία και το ερώτημα θα πρέπει να είναι τι ταιριάζει την ε, εκκίνηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, είτε μιλάμε για την αρχή του 2010 2000, όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε τους όρους για την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, είτε μιλάμε την καταστροφή της πρόσβασης σε αυτή τη χρηματοδότηση. Το θέμα είναι η ανάπτυξη κλάστερς γιατί οι επιχειρήσεις συνήθως δεν προκύπτουν από το μηδέν. Υπάρχουν και κλάστερς τα οποία συμβαίνουν. Πώς ε, διευκολύνουμε λοιπόν αυτή την ανάπτυξη, πώς συμμετέχουμε σε μια διαδικασία χωρίς να προσπαθήσουμε να εφεύρουμε κάτι το οποίο θα κολλήσει προκειμένου να μας οδηγήσει στην ανάπτυξη που χρειαζόμαστε για τη μείωση της ενεργείας στην Ευρώπη. Οι ορίζοντες για το 2020 λοιπόν. Η επιτυχία του προγράμματος εξαρτάται από τον ιδιωτικό τομέα και κατά πόσο θα αναπτυχθεί παράλληλα με τις γραμμές αυτές προκειμένου στο δημόσιο τομέα να δημιουργηθεί κάτι που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί εμπορικά. Και ελπίζουμε κάποιες από τις απαντήσεις να τις λάβουμε από τους εμπειρογνώμονές μας. Ο Πρόεδρος, ευχαριστούμε κυρία Σκίνερ. Θα δώσουμε ευθύς αμέσως το λόγο τώρα στον Πρόεδρο της ε, Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ. Μεγάλη μου τιμή που μιλώ για την βιομηχανική ηγεσία. Και θα είμαι σύντομος. Αντιμετωπίζουμε παγκόσμιες προκλήσεις. Οι πιο πολλές εξ αυτών είναι αρκετά συγκεκριμένες. Και θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε την εξέβρεση συγκεκριμένων λύσεων. Εκ παραλλήλου όμως υπάρχουν και κάποιες άλλες ε, προκλήσεις που δεν είναι συγκεκριμένες, να το θέσω έτσι. Η περιέργεια του ανθρώπινου είδους, η γνώση για το αύριο. Κοιτώντα τη βιομηχανική ηγεσία θα πρέπει να συνδυάσουμε αυτές τις δύο πτυχές με ένα πολύ σαφή τρόπο. Και εδώ στην εικόνα αυτή βλέπετε τη σχέση αυτή. Άρα από τη βασική έρευνα προς την αγορά από την ανακάλυψη στην κοινοτομία. Πρόκειται για μια ιστορία που ξεκινά από την περιέργεια και από τις παγκόσμιες προκλήσεις. Να σας δώσω κάποια παραδείγματα από την, ε, σε ό,τι αφορά την, ε, την αεροναυτική και την ε, διαστημική τεχνολογία. Σε ό,τι αφορά την παρατήρηση της γης, δορυφόρους και το, το Έχουμε βασικούς παράγοντες ε, επιτυχίας, η αναγνωρίση και η αποδοχή για την ανάγκη ευρωπαϊκής συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα, πολιτική θέληση για τη δημιουργία ανάλογων ευρωπαϊκών τομέων, δημιουργία και συνεχής ανάπτυξη κοινών ευρωπαϊκών χώρων και στρατηγικών έρευνας, εφαρμογή στρατηγικών με εναρμονισμένο τρόπο κατάλληλη χρηματοδότηση σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και ιδιωτικό επίπεδο που θα καλύπτει όλη την αλυσίδα έρευνας και η ύπαρξη συνεχούς αλυσίδας οικονομικής προστιθέμενης αξίας. Και αυτό μπορώ να σας το δείξω εδώ πέρα στο εικόνα αυτή. Χρειαζόμαστε λοιπόν στη διαδικασία καινοτομία σωστή χρηματοδότηση από την αρχή μέχρι τέλους, μέχρι να αναλάβει η βιομηχανία. Και αυτό δεν αποτελεί μόνο μία ιδέα, ιδιαίτερα για την ε, διαστημική τεχνολογία και για την αεροναυτική. Αποτελεί μία πραγματικότητα. Βλέπετε λοιπόν τα διάφορα βήματα τα οποία είναι πολύ ε, συγκεκριμένα ως προς τον ορισμό τους. Και επίσης είναι σαφής και ο ρόλος των εθνικών ε, κέντρων έρευνα, ο ρόλος της ε, Ακαδημίας, ο ρόλο των πανεπιστημίων. Επίπεδο ετοιμότητας τεχνολογίας 2 έως 3 σε συνεργασία με τον ακαδημαϊκό κόσμο. Επίπεδο 3 έως 5 και 6, ανάπτυξη νέων τεχνολογιών σε συνεργασία με τη βιομηχανία και φυσικά και η ε, εκπαίδευση των νεαρών εκπαιδευτών είναι πολύ σημαντικό θέμα. Έχουμε λοιπόν το Εθνικό Κέντρο Ερευνών που καλύπτει τον ε, θέμα της αεροναυτικής του διαστήματος, της ενέργειας και των μεταφορών και στην ε, αποστολή μας βλέπετε ότι στο κόκκινο τμήμα αναφέρεται να γευρεθεί το χάσμα μεταξύ της βασικής έρευνας και της ε, των κοινοτομικών εφαρμογών και μεταφορά της γνώσης και των αποτελεσμάτων έρευνας στην βιομηχανία. Για την αεροναυτική αυτό σημαίνει ότι δεν καλύπτουμε μόνο εθνικό τομέα, αλλά συνεργαζόμαστε σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο με διάφορους εταίρους και χαιρεόμαστε που και στο πρόγραμμα Horizon 2020 θα έχουμε την δυνατότητα συνεργασίας με τη ΣΥΠΑ. Κοιτώντας τώρα τι γίνεται στην αεροναυτική, είναι σαφής η ατζέντα μας για την στρατηγική Έχουμε πέντε στόχους. που καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα και οι διάφοροι παράγοντες για την επιτυχία της ατζέντα αυτής είναι να λάβουμε υπόψη το τι κάνουμε. Αναγνωρίζουμε την ε, αεροναυτική και τα συστήματα αεροπορικών μεταφορών ως ένα ε, ξεχωριστό σύστημα ευρωπαϊκής προτεραιότητας, να ορίσουμε τις απαιτήσει ε, ως προς την έρευνα για τις υποδομές, να διατηρήσουμε ε, τους μηχανισμούς υποστήριξης έρευνας και ανάπτυξης, να υπάρχει μια διαρκή ροή εκπαιδευμένων ανθρώπων και να υπάρχει μια αλυσίδα προμηθειών προκειμένου να, είναι, να υπάρχει συντονισμό σε, σε όλα τα επίπεδα. Να κοιτάξουμε τώρα σε ό,τι αφορά το διάστημα κάποιους ε, βασικούς ε, τομείς. Ε, εδώ έχουμε το θέμα των διαφόρων δορυφόρων, των κέντρων ελέγχου και διάφορων άλλων βιομηχανικών τομέων. Έχουμε και τα προγράμματα που ονομάζονται European Space Flagship Programs, όπως το Καλλιλέο για παράδειγμα. Το ερώτημα λοιπόν είναι κατά πόσο πρόκειται για πτυχέ του διαστήματος. Όχι, κοιτάξτε το ίδιο το, Γαλιλαίο, το πρόγραμμα Γαλιλαίο που ανταποκρίνεται σε ανάγκες της κοινωνίας. Για παράδειγμα, τη μείωση των επιπέδων η χορύπανση κοντά στα αεροδρόμια. Επίσης, διασφαλίζουμε την ε, ασφαλή χρήση των τρένων ε, χρησιμοποιώντας ένα σύστημα για την αποφυγή συγκρούσεων. Επίσης, το διάστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην επίλυση του ζητήματος της ενεργειακών αναγκών. Λαμβάνοντας υπόψη τη βιομάζα, γεωθερμικές, ε, ε, αιωλικές και άλλες πτυχές. Χρειάζεται επίσης και δημόσια ηγεσία η οποία θα πρέπει να οριστεί από τα διάφορα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία του Διαστήματος και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να καταλήξω λοιπόν τώρα σε κάποιες συστάσεις προκειμένου να διατηρηθεί και να κερδιθεί αυτή η βιομηχανική ηγεσία. Να υπάρχουν κατάλληλε στρατηγικέ, να υπάρχει κατάλληλη χρηματοδότηση σε όλα τα επίπεδα. Να υπάρχει χρηματοδότηση για το πρόγραμμα Horizon 2020, σύμφωνα με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2020, να υπάρχουν ε, επιτυχή μέσα για τα, όλα τα επίπεδα καινοτομίας, από τα μικρά, στα μεσαία και στα μεγάλα έργα. Να υπάρχουν ε, σωστά, σωστοί μηχανισμοί χρηματοδότησης. Και τέλος, να υποστηριχθεί και βιωσιμότητα της αλυσίδας. Να σας δείξω τι σημαίνει αυτό στην επόμενη διαφάνεια. Δεν φτάνει να κινούμαστε από τον ένα τομέα, από την αεροναυτική, για παράδειγμα, στο αεροπλάνο. Θα πρέπει να υπάρξει ε, πολλαπλή χρήση όλων των τομέων, για παράδειγμα, της ρομποτικής. Είναι πολύ σημαντική αυτή η διάδραση μεταξύ της παροχής κινήτρων και της ζήτησης. Το θέμα λοιπόν είναι πώς θα γίνει αυτή η διάδραση. Και η ιδέα φυσικά είναι να υπάρχει συνεργασία και μεταφορά μεταξύ των τομέων, να υπάρχει ένταξη όλων των τομέων που εμπλέκονται στην έρευνα και στην ανάπτυξη και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για να αποδεχτεί ότι για παράδειγμα, τα πορίσματα του ενός τομέα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε έναν άλλον. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε. Και τώρα, η Κέρα Ντεκάρα που είναι ε, General Manager, γενική Manager της, ε, της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης για το εμπόριο. Okay, thank you for the invitation. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Δύσκολο να κρατήσω την προσοχή σας να την, και να την σας εντυπωσιάσω μετά τα όσα είπε ο καθηγητής Λί που ήταν όλα αυτά τόσο συναρπαστικά και ενδιαφέροντα. Είμαι επομένως της IBAN ε, η, η manager και εκπροσωπούμε επομένω διάφορους ε, εμπόρους και επενδυτές. Θα προσπαθήσω να σας δώσω να καταλάβετε γιατί ο ρόλος μας είναι σημαντικός για την σημερινή μας προβληματική. Η φορέα μας συνενώνει πολλούς business angels. Τι θα πει αυτό, τι θα πει αυτό άγγελος της επιχείρησης. Υπάρχει ένας ορισμός, 27 χώρες συμμετέχουν σε αυτή την υπόθεση. Δεν το Είναι ένας ιδιώτης επενδυτής. Επενδύει τα χρήματά του. Και λαμβάνει μόνος του τις αποφάσεις. Αυτή είναι η διαφορά με άλλους επενδυτές. Εκείνοι, οι business angels, λαμβάνουν την τελική απόφαση για την επένδυση. Και εκτός από τα χρήματα είναι η επαφή με διευκολύνει την επαφή τόσο μεταξύ επιχείρησης δικτύου επιχειρήσεων και πελατών. 25 με 250.000 ευρώ είναι ο μέσος όρος ε, αυτών των επενδύσεων. ότι τα μεγάλα ποσά αφορούν δύο ή τρει τέτοιου business angels, τέτοιου Αγγέλου. Πρώτη για τι επιχειρήσει που ψάχνουν κεφάλαιο για να ξεκινήσουν τη δραστηριότητά τους. Προσφεύγουν λοιπόν σε αυτούς τους angels οι επιχειρήσεις και επίσης προσπαθούν να καλύψουν επομένω την έλλειψη ρευστότητα. Και αυτό πριν τη θέση εμπορία του προϊόντος που έχουν. Είναι η φάση κατά την οποία αναζητούν τις επενδύσεις οι επιχειρηματίες. Αυτό το λέμε equity gap. Τώρα έχουμε επομένω διάφορους φορείς και διαφορετικά, διαφορετικές κατηγορίες τέτοιων business angels. Επίσης μπορούμε να φτάσουμε από τις 20.000 μέχρι τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Και εδώ βλέπετε σε αυτή την διαφάνεια τα τα λόγο, τα λογότυπα διαφόρων χρηματοδοτουμένων εταιριών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ο ρόλο των Angels γιατί να βοηθούν τις επιχειρήσεις. Τώρα, τι, σε τι αποσκοπούν αυτοί οι Business Angels. Η, η ομάδα. αυτή που επενδύουν αυτοί που λαμβάνουν την επένδυση θα πρέπει να έχουν στρατηγική, θα πρέπει να έχουν κάποιο σχέδιο. Πολύ σημαντικός παράγον επίσης είναι θα υπάρχουν IP. 4 δις ευρώ σε 2.000 εταιρείε επενδύονται κάθε χρόνο. η οργάνωσή τους είναι σε δίκτυα, σε ομαδοποιούνται, σε τοπικό, τομεακό, περιφερειακό επίπεδο δρόν, και το, το μοντέλο στο οποίο βασίζονται ε, ποικίλει για να συμμετέχουν σε αυτές τις ενώσεις συνήθως πληρώνουν κάτι σαν συνδρομή. Επίσης υπάρχει και η φάση κατά την οποία γίνεται το ξεκαθάρισμα των προσφορών πριν γίνει η επένδυση. Εκπροσωπούμε επίσης και για κάποια ομοσπονδία τέτοιων δικτύων. Αυτά για να σας πω τι κάνουμε εδώ στις Βρυξέλλες. Τώρα μερικά αριθμητικά στοιχεία. Σας είπα ότι η αγορά είναι 3,5 δις ετησίως. Μας πλησιάζει αυτό, μου φαίνεται αυτό κοντά στα επίπεδα τα αμερικανικά. 2.000 και 300.000 όμως είναι οι business angels στην Αμερική. Ένα σε εμάς είναι επομένως 72.000. Τώρα, εδώ βλέπετε την κατανομή των επενδύσεων θυμίζει αυτά που είπε ο Ριγισλή. Βασικά έχουμε ε, την ε, ICT και κατόπιν έχουμε την κατάτμιση ανα αριθμό συμφωνιών. Να σας πω τώρα την εμπειρία της τελευταίας διετίας. Είχαμε το ICT, ήταν ένα πρόγραμμα, ούτω ώστε να παράσχει κάποιο είδους εκπαίδευση σε σχέση με το έκτο πρόγραμμα πλαίσιο. Θέλαμε να βρούμε επομένω κάποιες εταιρείες, 20.000 εταιρείες έπρεπε να... 20.000 ερευνητικά προγράμματα λέει τώρα η μιλήτρια, που έλαβαν χρηματοδότηση στα πλαίσια του προγράμματος πλαισίου και αυτούς θα να τους φέρνουμε σε επαφή με τους επενδυτές, να τους δώσουμε επομένω την ε, ευκαιρία για επενδύσεις, ε, κατάρτιση και την ευκαιρία επομένω να μπορέσουν να παρουσιάσουν το, το πρόγραμμα στους επενδυτές για δύο, μισή χρόνια κράτησε αυτή, αυτό το αυτή η δουλειά σε όλη την Ευρώπη. Ε, ψάξαμε, καλέσαμε ε, ερευνητέ ε, από τα πανεπιστήμια να παρουσιάσουν το πρόγραμμά τους. Τώρα σχεδόν ολοκληρώθηκε αυτή μας η προσπάθεια. Εξασφαλίσαμε χρηματοδότηση, έχουμε διατυπώσει κάποιες συστάσεις για το τι πρέπει να βελτιωθεί, στο πώς αξιολογούνται αυτά τα ερευνητικά προγράμματα. Το πιο σημαντικό μας συμπέρασμα είναι ότι λίγα μόνο από αυτά τα προγράμματα φτάνουν στη φάση της ε, εμπορίας. Καμιά φορά είναι μεγάλος ο κίνδυνος, καμιά φορά δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδρομή του προγράμματος. Οπότε ε, έχουμε αυτόν τον κατάλογο των επενδυτών. Απευθυνθήκαμε σε όλους. Ήταν δύσκολο να τους πείσουμε να έρθουν και να συναντήσουν και να τους πείσει να έρθουν επομένως ε, και οι ερευνητές όλοι εδώ και να παρουσιάσουν το έργο τους στους επενδυτές. Δεν υπάρχουν και τόσες περιπτώσεις όπου έρχονται οι ερευνητές να τα παρουσιάσουν τους γεώτες. Οπότε είναι δύσκολο οι επενδυτές να μπορέσουν να δουν το τι περιέχει το, κάθε πρόγραμμα, κάθε φάκελος. Επομένως, γι' αυτό αξίζει αυτό το οποίο κάναμε. Και επομένως έτσι συμβάλλουμε σε αυτά τα ε, προγράμματα. Βεβαίως είναι και το θέμα των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Να σας πω τώρα, τι συστάσεις κάναμε προς τους ε, policy makers. Αυτό το οποίο είπε και ο Πρώτα πρώτα. Να αυξηθεί το capacity building. Θα πρέπει ομένως οι επενδυτές να συμμετάσχουν σε κάποιες φάσεις του προγράμματος. Πρώτα πρώτα η Επιτροπή αξιολογεί το πρόγραμμα. Κατόπιν ο επενδυτής και αυτός θα πρέπει να αξιολογήσει. πρέπει να εκπαιδεύσει τον επιχειρηματία, αλλά από την αρχή και όχι μόνο στην ύστερη φάση. Έτσι θα προλανθεί το έδαφος. Για να γίνει καλύτερη η διαδρομή του προγράμματος από την έρευνα μέχρι την αγορά. Αυτός πρέπει να είναι ο, ο ρόλος τους σε όλη αυτή την διαδρομή. Επίσης, προτείναμε τη μερία κάποιων ταμείων και έχουμε κάποιες συστάσεις για διασυνοριακές δραστηριότητες και έχουμε μόνος, αυτό το ταμείο τις, ε, τόν τον για, για τις ε, επενδύσεις με τους business angels. Και επίσης είπαμε ότι αυτό που ανέφερε ο Ζόμπι, πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν και φορολογικά κίνητρα. Υπάρχουν στοιχεία που κατακρίνουν ότι όποτε υπήρχαν τέτοια κίνητρα, και για τις καινοτόμες εταιρείε, αλλά και οι επενδυτές να έχουν φορολογικά κίνητρα. Αυτό έφερε πάρα πολύ θετικά αποτελέσματα. Αυτό έγινε όπως θα ξέρετε και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τέτοιε συμβουλέ δώσαμε επομένω και είπαμε ότι θα θέλουμε να τονώσουμε έτσι την αγορά ενώ του 2020. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η κυρία Γκινέα θα λάβει τώρα το λόγο. Ο κύριος Φούλβιο Ουτζέρη δεν μπόρεσε να παρευρεθεί, Ζητήσει γνώμη. Θα τον εκπροσωπήσω εγώ και θα ε, παρουσιάσω κάποιες απόψεις για την Ευρωπαϊκή Χημική Βιομηχανία. Είναι υψηλές ε, οι φιλοδοξίες ε, που τίθενται τώρα. Υπάρχουν πάρα πολλές προτάσεις επίσης για τη μείωση της, των ρήπων της κατανάλωσης ενέργειας. Όλα αυτά χρειάζονται και συνεπάγονται υψηλές προσδοκίες. Είναι σαφές ότι για να επιτευχθούν οι στόχοι η καινοτομία είναι ένα εργαλείο ουσιαστικό. Όταν λέω καινοτομία δεν μιλάω μόνο για νέες επιχειρήσεις, αλλά μιλάω και για την αναζωογόνηση της βιομηχανίας μας όλων των κλάδων της βιομηχανίας και της κοινωνίας. Πρέπει λοιπόν το μέσο αυτό να προοικοδοτηθεί με αυτά που χρειάζεται το Horizon 2020. Χρειάζονται ισχυρά πολιτικά μηνύματα και οικονομικά, αλλά και θα πρέπει να τεθεί ένα πλαίσιο. Τα θεσμικά όργανα και όλοι θα πρέπει να δώσουν μάχη για να προαχθεί η οικονομία και η ανταγωνιστικότητα. Συμφωνούμε με την απλοποίηση. Είναι σημαντικό να συνεχιστεί και να βελτιωθεί η κατάσταση εδώ. Δεν ε, ε, μιλάμε μόνο για την προώθηση των ε, προϊόντων. Χρειάζεται συντονισμός γενικότερος και η Επίτροπος μίλησε για τη συνεργασία των τριών πυλώνων. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Θα δούμε πώς θα λειτουργήσει στην πράξη όμως. Ένα πρακτικό μέσο είναι η χρήση της υπάρχουσας ευρωπαϊκής τεχνολογικής πλατφόρμας που μπορεί να βοηθήσει και θέματα καινοτομίας. Κάτι που πετύχαμε με το Horizon 2020 e είναι ότι ίσως κάναμε επιτέλους τη διάκριση μεταξύ έρευνας και καινοτομίας. Γιατί δεν είναι τα ίδια αυτά τα δύο. Η καινοτομία είναι να πάμε τα ερευνητικά αποτελέσματα στην αγορά. Ο πυλώνας της βιομηχανικής, η θύνουσας θέσης υπογραμμίζει τον παράγοντα της θέσης στην αγορά. Εδώ χρειάζεται αναβάθμιση και μια ουσιαστική ε, πολιτική ε, για την εμπορική εφαρμογή. Χρειάζονται κανόνες σαφέστεροι, κανόνες που να μπορούν να εφαρμόζονται στη διαχείριση Έχουμε θέσει στόχους για τη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Χρειάζεται όμως να διευκρινίσουμε τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουμε για να πετύχουμε το στόχο. Καλό είναι να δοθούν κίνητρα, όχι μόνο στις καινοτόμες, όπως λέμε, επιχειρήσεις, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μην ξεχνάμε και τις παραδοσιακές. Γιατί οι παραδοσιακές ποιες είναι. Είναι οι συνήθεις είναι η κλάδη της παραγωγής μας, η κλασική που μπορεί και αυτοί να καινοτομούν και αποτελούν και τη βάση των οικονομιών μας. Μπορούν να αποφέρουν τεράστια ωφέλη στην Ευρώπη, ώστε η Ευρώπη να ωφεληθεί σε ανταγωνιστικό επίπεδο σε σχέση με τις άλλες περιοχές του κόσμου. Χρειάζεται ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ μικρομεσαίων και μεγαλύτερων επιχειρήσεων. Και κάποιος πριν είπε ότι όλα αυτά δεν γίνονται έτσι εκ του μηδενός. Ένα πλεονέκτημα της Ευρώπης είναι αυτή, αυτό το ομαλό ε, δίκτυο που υπάρχει μεταξύ των επιχειρήσεων. Είναι κοντά η μία στην άλλη, συνεργάζονται και υπάρχει και ένα γεωγραφικό πλεονέκτημα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, γιατί έτσι μπορεί να οικοδομήσει η μία πάνω στις δεξιότητες της άλλης. Τώρα, για τη βιομηχανική ηθήνουσα θέση θα πρέπει να αξιολογήσω με το πρόγραμμα όχι μόνο με επιστημονικά κριτήρια, αλλά και με βάση τον αντίκτυπο στην αγορά και κάποια ειδικότερα στοιχεία και κριτήρια αξιολόγησης πρέπει να αναπτυχθούν. Θα ήταν ευπρόσδεκτο αν οι αξιολογητές ε, από βιομηχανικούς τομείς ε, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν γιατί και εκείνοι έχουν μια ειδική συμβολή. Επίσης, είναι πολύ καλή η πρόταση για επιστροφή του 100% του κόστους, ε, αλλά Καμιά, ε, το, η, ε, η, πρόβλεψη ε, για 100% λογιστική καταχώρηση του κόστους είναι κάπως δύσκολο για τις επιχειρήσεις. Επίσης, Επίση, καλό είναι και αυτό το, η πρόβλεψη για το έμεσο κόστος μέχρι 40% γιατί είναι πάνω από 20% οι περισσότερες. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να υπάρξουν συμπράξεις σε δημοσίου ιδιωτικού τομέα ε, και, καλή είναι και ε, καλές είναι και οι κοινέ προγραμματικές ε, πρωτοβουλίες. Αλλά ο διάβολος κρύβεται στη λεπτομέρεια. Πρέπει να δούμε πώς θα λειτουργήσουν όλα αυτά. Είναι σημαντικά εργαλεία ανάπτυξης. Οι ΣΔΙΤ, οι συμπράξεις δημοσίου ιδιωτικού τομέα, θα πρέπει να εξετάζουν θέματα καινοτομιών και χρειάζεται να προσαρμοστούν Ω προ την καινοτομία. Υπάρχει ένα, υπήρχε ένα πρόγραμμα πλαίσιο που ήταν 100% αφιερωμένο στην έρευνα. Η καινοτομία όμως πρέπει να ε, συμπεριληφθεί ακόμη περισσότερο υπόψη μέσα από καινούρια μέσα. Επίσης, οι ΣΔΙΤ είναι σημαντικές γιατί εκφράζουν κοινή δέσμευση για ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Είναι κοντά στην αγορά. Μπορεί να επιφέρουν εκείνη την κρίσιμη μάζα που χρειαζόμαστε. Η συμμετοχή των κρατών μελών είναι σημαντικό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορεί να συντονίζει τις δραστηριότητες των κρατών μελών για να ε, υπάρχουν σωστοί ορισμοί των κοινών προγραμματικών πρωτοβουλειών. Να πω επίσης κάτι για τον τομέα το, τον χημικό και να κάνω και κάποιες προτάσεις σε σχέση με αυτά που μπορούμε εμείς να κάνουμε, όχι μόνο τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ότι μπορεί και ο κλάδος μας να κάνει, γιατί δεν μιλάμε εδώ μόνο για λεφτά, Είμαι βέβαιη ότι οι εταιρείε μας θα συνεχίσουν να είναι καινοτόμες και θα αναπτυχθούν εξαιρετικά σε όλο τον κόσμο. Αυτό που χρειάζεται όμως είναι να έρθει νέα αξία στην Ευρώπη, προστιθέμενη αξία, αφού ανταγωνιζόμαστε άλλες περιοχές του κόσμου. Χρειάζεται λοιπόν ένα μοντέλο καινοτομία το οποίο θα ταιριάζει στην Ευρώπη. Ένα μοντέλο καινοτομία που θα στηρίζεται στα πλεονεκτήματα της Ευρώπης, αυτά που έχουμε εμείς εδώ, που λαμβάνει υπόψη την αλυσίδα της αξίας και πρέπει να διαφοροποιήσω μεταξύ αλυσίδας καινοτομίας και αλυσίδα αξίας. Μπορείτε να μου πείτε ότι όλα αυτά είναι τώρα σημασιολογικά και ε, σημειολογία. Αλλά υπάρχει διαφορά μεταξύ έρευνας και αγοράς και η αλυσίδα της αξίας είναι από τον προμηθευτή των υλικών μέχρι τον τελικό χρήστη του προϊόντος καλό είναι να χρησιμοποιήσουμε αυτή την αξιακή αλυσίδα, αν θέλετε, αυτό το μοντέλο αλυσίδας αξίας που έχουμε στην Ευρώπη, επειδή είναι έτσι η γεωγραφική εγκύτητα των διαφόρων τομέων στην Ευρώπη. Ε, έτσι θα μπορέσουμε να κάνουμε τα άλματα που πρέπει να κάνουμε στην Ευρώπη. Μέσα από αυτό το μοντέλο θα μπορούσαμε να δώσουμε κίνητρα, αν θέλετε, ε, ώστε να λειτουργήσει στα διάφορα στάδια της αυτή η αλυσίδα της αξίας. Οι διάφοροι τομείς κατά μήκο της αλυσίδας της αξίας θα ε, ε, υποστούν σε διαδικασίες όθησης και έλξης προς νέες τεχνολογίες, προς νέα προϊόντα, προς την αναζωογόνηση του τομέα τους κλπ. κλπ. Μέσα από αυτό το πρίσμα η ευρωπαϊκή χημική βιομηχανία ως ευρωπαϊκός τομέας για πρώτη φορά βγαίνει με πρόθεση της καινοτομίας, όθηση, γιατί πιστεύουμε ότι μπορούμε να είμαστε πολύ σημαντικός εταίρος στις διάφορες συμπράξεις για την καινοτομία που τώρα βλέπουν το φως της μέρας είτε στο, στα νέα υλικά ή στην, ε, στις έξυπνες πόλεις ή στην ενεργειακή απόδοση κλπ. Θα ήθελα τέλος να πω ότι τώρα στην Ευρώπη είμαστε σε, μια, σε ένα δίλημα θα πρέπει ε, να ε, πιέσουμε την καινοτομία και σε οικονομικό επίπεδο μέσα από τη χρηματοδότηση αλλά και μέσα από μια καλά ε, καταρτισμένη στρατηγική. Πρέπει να δώσουμε ελπίδα και όνειρα γιατί η καινοτομία αφορά την επίλυση των προβλημάτων, αλλά σημαίνει και δημιουργία νέων οραμάτων, να αξιοποιήσουμε περιοχές που ακόμα δεν έχουν χαρτογραφηθεί. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Και η κυρία Φόρτα έχει το λόγο. Thank you. It's a question Thank Σας ευχαριστώ για την φανταστική σας ε, παρουσίαση. Μία ερώτηση για το επιχειρηματικά κεφάλαια. Στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε τα διευθυντικά ταμεία που χρησιμοποιούνται για τη συγχρηματοδότηση επιχειρηματικών κεφαλαίων. Όχι όμως συγκεκριμένα για να βοηθηθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις των οποίων ε, χρηματοδοτείται η έρευνα μέσω ευρωπαϊκών επιδοτήσεων. Θα βοηθούσε, θεωρείτε, να χρησιμοποιηθούν κάποιοι πόροι για αυτό συγκεκριμένα, γιατί δεν είναι όλοι, δεν θέλουν όλοι οι ερευνητέ εμπορευματοποίηση των σκέψεων και των ιδεών τους, αλλά σαφώς υπάρχει ένα χάσμα σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην αγορά των επιχειρήσεων αυτών. Άρα, μήπως θα ήταν χρήσιμο να δαπανηθούν κάποιοι από τους πόρους που προορίζονται για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για ένα ταμείο το οποίο θα συγχρηματοδοτήσει τα επιχειρηματικά κεφάλαια μέσω των Business Angels. Ευχαριστώ. Η κυρία Τόμψεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ έχω μια ερώτηση την οποία θα πρέπει να συζητήσουμε επί της αρχής. Πώς ορίζουμε τη βιομηχανία. Στα αγγλικά η βιομηχανία εννοεί όλες τις βιομηχανίες, όλους τους κλάδους, γιατί στα γερμανικά αυτό εμπεριέχει μόνο τους βιομηχανικούς παραγωγικούς κλάδους. Νομίζω ότι θα πρέπει να ορίσουμε ότι δεν μιλάμε μόνο στην απτή οικονομία. Γιατί μας είπε ο Αμερικάνο προσκεκλημένο μας σήμερα ότι 40% των θέσεων εργασίας στον τομέα του ICT είναι στον τομέα EPS. Αλλά, για παράδειγμα, στα computer games, που είμαστε πολύ καλοί στην Βόρεια Ευρώπη. Πίτερ, λιγότερο από 15% απασχολείται στην βιομηχανία. Εσείς έχετε μια δημιουργική βιομηχανία της μουσικής pop, για παράδειγμα, στην ε, Αγγλία. Κάθε φορά που είμαστε εδώ στην αίθουσα ακούμε για το διάστημα, για τη χημική βιομηχανία. Το σέβομαι και το πιστεύω ότι πρέπει να δραστηριοποιηθούμε στους τομείς αυτούς, αλλά θα πρέπει να ακούσουμε και το πώς ε, θα υπάρξει έρευνα για την απτή οικονομία, για τον τουρισμό στη Μαγιόρκα, γιατί σας διαβεβαιώ ότι θα πρέπει να ζήσουμε τον τουρισμό στο μέλλον στην ε, Ευρώπη. Είναι δημογραφικό το θέμα. Θα πρέπει λοιπόν να ορίσουμε το τι περιλαμβάνει ο όρος τουρισμός και πώς θα βελτιωθεί η απτή οικονομία, πώς θα ενταχθεί στο πρόγραμμα πλαίσιο. Ευχαριστώ πολύ. η κυρία Κόβιτς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε. Η αλήθεια είναι ότι το είναι πάρα πολύ συναρπαστικά και μου, μου, έδωσε την αφορμή να σκεφτώ, να προβληματιστώ. Ο κύριο Βέρνερ μέσα μα είπε, διότι κατά αυτόν τον τρόπο έχει καταστεί σαφέ ότι η διαδικασία της καινοτομία χρειάζεται μία μακρόπνοη, πολύ μακρόπνοη διαδικασία προγραμματισμού. Γιατί μόνο κατά αυτόν τον τρόπο είναι δυνατόν να καλυφθούν όλες οι περιπτώσει, όλε οι τάσει. Έχω επομένως για εκείνον μία ερώτηση. Πέστε μας παρακαλώ, πώς μπορούμε να πείσουμε τον ε, αγοραστή για να αγοράσει κάτι το οποίο είναι πολύ προηγμένο τεχνολογικά. Γιατί μιλάμε για τέτοιου είδους πάρα πολύ απαιτητικά ούτως υπήν προϊόντα. Τώρα για την κυρία ε, Κάρο έχω μια ερώτηση. Πρόκειται για κάτι άλλο. Πρόκειται για το ότι θα πρέπει να παρουσιάσουμε για τους, ε, για αυτούς τους αγγέλους των επιχειρήσεων κάποια συγκεκριμένα στοιχεία. Ε, πολλές φορές δεν μπορούν οι ίδιοι να κάνουν την έρευνα, θα πρέπει σε αυτό να το κάνουν στις τους τα πανεπιστήμια. Τα πανεπιστήμια να κάνουν την έρευνα για ένα προϊόν, για μια υπηρεσία. Αυτό επομένως χρειάζεται να γίνει. Πολλές φορές επίσης οι ερευνητές ε, πρέπει να, να, να, να, άρουν αυτή την έλλειψη, θα πρέπει να, αυτό το κενό να το γεφυρώσουν, γιατί καθόλου τον τρόπο μπορεί τελικά να τεθεί σε εμπορία ένα συγκεκριμένο προϊόν. Μετά έχουμε το venture capital, το κεφάλαιο επιχειρηματικού κινδύνου, το οποίο θα πρέπει επίσης να το, το αγκαλιάσουν ε, οι φορείς που πρέπει και έτσι να πιστούν ε, για το ότι αξίζει να ασχοληθούν ε, οι επενδυτές με κάποιο συγκεκριμένο προϊόν. Κύριε Βόρνερ, παρακαλούμε μια σύντομη απάντηση δώστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα πώς ορίζεται ο όρος βιομηχανία. Γερμανός είμαι, ξέρετε. Δεν πρόκειται να πω ότι η βιομηχανία είναι μόνο η κατασκευή κάποιου προϊόντος. Για μένα είναι ε, μπορεί να καλυφθεί και η ιατρική, μπορεί να καλυφθεί και η γεωργία. Δεύτερον, πώ μπορούμε να πάρουμε κάποιε εγγύσει για το ότι κάποιο προϊόν θα φτάσει στην αγορά. Έχετε δίκιο 100%. Συνήθω οι ερευνητέ δεν είναι εκείνοι οι οποίοι ε, κάνουν τι απαραίτητε δημόσιε σχέσει προ Άρα θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την ανταγωνιστικότητα του προϊόντου, τον ενελκυστικό το προϊόν, η λειτουργία του προϊόντος είναι σημαντική και στην αεροναυπηγική, ξέρετε, είναι επίση. Ε, είναι επίσης πολύ σημαντικό το να υπάρχει ε, η αναγκαία ετοιμότητα, να υπάρχει πιστοποίηση του προϊόντος και αυτό επίσης γίνεται και σε άλλους ε, τομείς. Παράδειγμα, κοιτάξτε τι γίνεται με τα κινητά τηλέφωνα. Λένε ότι πουλούνται ακόμα και αν δεν δουλεύουν. Να, επομένως, ε, ένα παράδειγμα του τι πάει να πει δημόσιες σχέσεις. Χρειάζεται έτσι ένα ελκυστικό καλό προϊόν, ε, που να λειτουργεί και επίσης ε, και οι νέοι επιχειρηματίες που ξεκινάνε μια επιχείρηση χρειάζεται να έχουν και ε, κάποιους δημόσιες σχέσεις. Ευχαριστούμε πολύ, λέει Πρόεδρος. Κυρία Κιάρα Ντεκάρα, τώρα το λόγο. Δύο λεπτάκια. Ναι. Για τις ΜΜΕ ήταν η πρώτη ερώτηση. Συμφωνώ 100%. Ο ρόλος τους είναι πολύ σημαντικός. και για την ε, καινοτομία. Αυτό που είπαμε όσον αφορά για αυτό το, το, το φαινόμενο του καταράκτη που είπε ο κύριος Ένα ολόκληρο σύστημα εδώ πέρα αποδίδει την εικόνα και αυτό θα πρέπει να προσέξουμε. Βλέπουμε επίσης εδώ την εμπλοκή και των μεγάλων εταιριών στις πρώτες φάσεις. Βεβαίω, πολλές φορές θέλουν να κάνουν τις δικές τους εταιρείες οι επενδυτές. Όμως χρειάζεται υποστήριξη των ΜΜΕ που είναι οι καινοτόμες. Και εκείνες ελκύουν τους περισσότερους επενδυτές και από άλλες χώρες και διασυνοριακά. Δεύτερη ερώτηση. Συμφωνώ για αυτό που είπατε για τους ερευνητέ. Θα πρέπει να υπάρχουν δεξιότητες, ο χρόνος δεν υπάρχει πάντοτε. Από την αρχή της ανάπτυξης ενός προϊόντος θα πρέπει να υπάρχει κάποιος ειδικό στο μάρκετινγκ στην ομάδα. να υπάρχει και μια στρατηγική που να εκπονήσουν με κάποιον ε, έμπειρο επιχειρηματία ή έναν ε, έμπειρο ε, άγγελο επιχειρήσεων. Λορεντάνα Κινέα. Thank you. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να μιλήσω για τη βιομηχανική παραγωγή. την παραγωγή προϊόντων. Για να δούμε τα πλεονεκτήματα της Ευρώπης εδώ. Μπορεί να παρακολουθήσει τους ανταγωνιστές της στην πληροφορία, την επικοινωνία, σε αυτές τις τεχνολογίες. Έχουμε κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να προασπίσουμε τα στρατηγικά συμφέροντα της Ευρώπης. Δεν το έχουμε εξαντλήσει το θέμα, πιστεύω. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ε, τους ηλιακούς συλλέκτες Έχουμε κάνει όλη την έρευνα και την ανάπτυξη εμεί στην Ευρώπη. Όλοι όμω κατασκευάζονται στην Κίνα και από εκεί τους αγοράζουμε. Ε, πρέπει λοιπόν να επικεντρωθούμε στις ανάγκες της Ευρώπης, τα επιτεύγματα της Ευρώπης με τα μέσα που διαθέτουμε. Δεν μπορούμε βέβαια να κάνουμε τις επενδύσεις που κάνει η Αμερική η Κίνα στην έρευνα και την καινοτομία, ούτε έχουμε την ίδια δομή διακυβέρνησης όπως αυτή που τρέχουν γρήγορα και οι διαδικασίες όταν θέλουν είναι ταχύτατες. Αυτό πρέπει να το δεχτούμε, να συμβιβαστούμε με αυτό και να το αντιμετωπίσουμε βέβαια και εμείς όπως μπορούμε. Η κυρία Γκράτσια Καρβάλιο. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω τους ομιλητές. Κράτησα πολλές σημειώσεις των συστάσεων που έκαναν. Εγώ θέλω να αναφερθώ σε αυτό που είπε η συνάδελφος Ρίτα Τόμσον. Ο ορισμός της βιομηχανίας πρέπει να είναι κατά ανάγκη γενικός. Θυμίζω όμως ότι το ICT, οι τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνία, συμπεριλαμβάνονται τις προτάσει τη Κομισιόν. Στη βιομηχανική θύνουσα ε, θέση που επιδιώκουμε, η ICT είναι πολύ σημαντικές. Βέβαια, θα πρέπει να διευρυνθούμε και σε άλλες εφαρμογές και σε άλλους τομείς. Και επίσης η έρευνα από κάτω προς τα πάνω δεν πρέπει να περιορίζεται στον πρώτο πυλώνα της αριστείας, πρέπει να διευρυνθεί και στην κοινωνική πρόκληση και στην ε, ε, βιομηχανική ηθήνουσα θέση και θα διευρύνουμε περισσότερο τον ορισμό της βιομηχανίας σε σχέση με τον ορισμό που δίνει η Κομισιόν. Οπότε συμφωνώ σε τελευταία ανάλυση με την πρόταση τη δική σας. Ευχαριστώ, κύριο Σκίνερ. Ευχαριστώ. Να απαντήσω σε αυτό που είπε η Βίκη Φόρντ. Το Ηνωμένο Βασίλειο είχε περιφερειακούς αναπτυξιακούς φορείς μέχρι που αποδομήθηκαν από την τωρινή κυβέρνηση και έχουν τώρα περιφερειακά κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου. Τώρα χρειάζεται να επαναλάβουμε αυτό που είχαμε κάνει και να ξαναγυρίσουμε στους περιφερειακούς αναπτυξιακούς φορείς και να δημιουργήσουμε μια αντίστοιχη υποδομή σε όλη την Ευρώπη. Γιατί αυτό που το είναι καλό σε περιφερειακό επίπεδο είναι καλό και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό. Ε, ε, βεβαίως είναι πολύ ε, σημαντικό να έχουμε apps. Πρέπει να εξετάσουμε όμως από πού θα προέλθουν από τις μικρές επιχειρήσεις, γιατί εκεί γίνονται οι εφευρέσεις και τώρα ε, είναι σε αυτή τη φάση. Ε, πρέπει επίσης να δούμε και τους τομείς προϊόντων και την ομάδα στόχου που Τώρα για το κεφάλαιο κινδύνου. Βεβαίως πρέπει να περάσουμε το μήνυμα για το κεφάλαιο κινδύνου. Αλλά εδώ στην Ευρώπη έχουμε πολύ περιορισμένο πεδίο εφαρμογής ε, για, τις, ε, ε, για τα επενδυτικά κεφάλαια. Επίσης, έχουμε περιορισμούς λόγω της ρευστότητας των τραπεζών και από την άλλη πλευρά λέμε «Α, οι ΜΜΕ έχουν αυτές και αυτές τις κεφαλαιακές ανάγκες». Δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Δεν μπορεί δηλαδή να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Στην Αμερική βλέπουμε ε, ότι τώρα ε, δημιουργούνται τράπεζες που είναι προσανατολισμένες ε, στις αναπτυξιακές ανάγκες των επιχειρήσεων. Αν δεν κάνουμε κι εμείς κάτι παρόμοιο, δεν πρόκειται να πάμε μακριά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές και σας, σας ευχαριστώ. Τελειώσαμε και αυτή την τρίτη συνεδρία και προχωρούμε ε, στην τέταρτη και τελευταία. Έχουμε και μια καθυστέρηση περίπου 20 λεπτά. Έχουμε καλύψει ε, μεγάλο κομμάτι της καθυστέρησης πάντως.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 αρχίζουμε επομένω στο τελευταίο τμήμα της ε, συνεδρίασης. Ε, Βεβαίω και έχει αρχίσει να βγαίνει η κούραση, αλλά θα προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε την προσοχή μας και να ακούσουμε προσεκτικά τους ομιλητές. Και τώρα, κύριε Έλερ, εισαγωγή. Πρόεδρε, συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, τα θέματα είναι πολύ ενδιαφέροντα γιατί πρόκειται για λεφτά. Θα μιλήσουμε για χρήματα. Θα ήθελα στο σημείο αυτό, στο τελευταίο τμήμα της ακροασής μας, ε, για το θέμα να μιλήσουμε για το θέμα των κανόνων συμμετοχής και καλωσορίζω ε, τους ε, παράγοντας που εμπλέκονται στο θέμα αυτό δεν χρειάζεται να σας εξηγήσω πόσο μεγάλες είναι οι προκλήσεις στο θέμα των κανόνων συμμετοχής σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στο πρόγραμμα πλαίσιο και το θέμα της απλοποίησης. Διαβάσατε τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μπορείτε να κρίνετε κατά πόσο οι αλλαγές θα μας ε, διευκολύνουν ή θα μας ε, κάνουν πιο δύσκολη τη ζωή. Νομίζω ότι το πάνελ αυτό θα εστιαστεί κυρίως σε θέματα κανόνων συμμετοχή. Νομίζω ότι ε, ως προς την αρχή, σε θέματα των κανόνων και απλοποίησης, βρισκόμαστε πριν από ένα μεγάλο άλμα γιατί πριν από δύο-τρία προγράμματα δημιούργηκε μία σοβαρή απόπειρα ε, πιο ελκυστικής διαμόρφωσης του προγράμματος προκειμένου να καταστεί και πιο ανταγωνιστικό σε διεθνές επίπεδο. Νομίζω ότι πριν αρχίσουμε να μιλάμε για τα προβλήματα, ότι αυτό ήταν ένα καθοριστικό βήμα και θα πρέπει να είναι καθοριστικό βήμα και για την ελκυστικότητα του προγράμματος Horizon 2020. Νομίζω ότι όλες οι ομάδες το υποστηρίζουν αυτό. Μειώσαμε τις ε, προδιαγραφές για το ωράρια εργασίας, επίσης ε, και το κόστος, το φορολογία ε, προστιθέμενης αξίας ε, αναγνωρίζεται ως μέσο και παρόλα αυτά, πέρα από τα επιτεύγματα αυτά, εξακολουθούν να υπάρχουν κάποια σημαντικά σημεία τα οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερο πρόβλημα, τα οποία τους επόμενους μήνες θα πρέπει να τα συζητήσουμε με το Συμβούλιο και με την Επιτροπή. Το πιο αμφιλεγόμενο είναι το ενιαίο ε, μοντέλο επιστροφής κόστους. Υπάρχουν ε, δύο συμβούλια. 100% καταρχάς ε, ποσοστό επιστροφής ή 70% για παράδειγμα της 100% και 20% για προγράμματα ερευνών για τα πανεπιστημιακά προγράμματα ε, είναι 100% εκάλυψη. Αλλά μειονέκτημα τέτοιας ρύθμισης είναι το έμεσο κόστος, το οποίο είναι πολύ υψηλό, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά μη πανεπιστημιακούς φορείς. Θα πρέπει να βρούμε μια ενδιάμεση λύση και για τη συζήτηση κάναμε κάποιες καλές προτάσεις θα μπορούσαμε να φανταστούμε, για παράδειγμα, μία λύση ενός μοντέλου επιστροφής του πλήρους κόστους ε, για κάποιους φορείς με δυνατότητα opt-out, αλλά το θέμα δεν είναι, ότι δεν πρόκειται μόνο για ένα συμβιβασμό που θα μας ικανοποιήσει όλους, αλλά για κάτι το οποίο δεν θα περιπλέξει τη διαδικασία, την ε, περαιτέρω διαδικασία του προγράμματος. Τελευταίο σημείο που θα ήθελα να αναφέρω είναι το όλο ζήτημα των διαφορών ε, ποσοστών ε, ενίσχυσης για διάφορες ε, κατηγορίες δραστηριοτήτων. Θα πρέπει να δούμε πώς θα γίνει αυτή η πρακτική διάκριση. Να δούμε λοιπόν πού σταματάει η έρευνα και πού ξεκινάει η κοινοτομία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το εγχείρημα αυτό και πολλοί κίνδυνοι ενέχονται. Αλλά ασφαλώς θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι κινούμαστε και σε ένα διεθνές προσκήνιο. Δηλαδή έχουμε μια απόφαση του ΠΟΕ για την Boeing όπου αναμένουμε ότι οι Αμερικάνοι και οι διεθνεί σκηνή θα παρακολουθήσουν με προσοχή ποιο θα είναι το καθεστώς που θα επικρατήσει για την καινοτομία. Γιατί τα πράγματα είναι αρκετά σαφή σε ό,τι αφορά την έρευνα στο θέμα της καινοτομία. Θα πρέπει να διατυπωθεί ξεκάθαρα όχι μόνο η διάταξη του προγράμματος, αλλά να δούμε και τι γίνεται από πλευράς επιδοτήσεων προκειμένου να υπερασπίσουμε τη θέση μας και στον ΠΟΕ. Χαίρομαι ιδιαίτερα λοιπόν που σήμερα έχουμε μαζί μας ε, μια σειρά φορέων από πανεπιστήμια, από τον ε, τομέα έρευνας εκτός των πανεπιστημίων και από ένα κλασικό βιομηχανικό τομέα της αεροναυτικής ο κύριος Giovanni Μπερτολόνε, πρόεδρος της Επιτροπής ε, του ASD, ο κύριος Γιάν Μέγγελερς, ο οποίος είναι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Οργανώσεων Έρευνας και Τεχνολογίας, ERTO, και τέλος η Dr. Jennifer Barnes, η οποία είναι αντιπρόεδρος για την Διεθνή Στρατηγική του Πανεπιστημίου του Cambridge που προσκλήθηκε στα πλαίσια της ομάδας Russell. Να ξεκινήσουμε πάρα αυτά γιατί έχουμε χάσει πάρα πολύ χρόνο και δίνει το λόγο κατευθείαν στον κύριο Τζιωβάνι Μπερτολόνα. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Έλλαρ, κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι, είναι ιδιαίτερη η χαρά μου που βρίσκομαι εδώ σήμερα το απόγευμα εξ ονόματος των κλάδων αεροδιαστημικής και άμυνας στην Ευρώπη. Βέβαια μετά την ε, παρουσίαση του καθηγητή Μπάρτον Λί έπαθα κρίση ταυτότητας γιατί λέω εμείς τι είμαστε, είμαστε βιομηχανίες στις μεταφορές ή στο ε, λογισμικό ή πώς μπορούμε να δεχτούμε ότι οι βιντεοδιασκέψεις ε, μειώνουν το, το χρόνο μεταφοράς ε, των εργαζομένων ή ε, πώς μπορούμε να συμπεριλάβουμε στον κλάδο μας απομακρυσμένες περιοχές. Είναι πολλά τα θέματα. Μετά ησύχασα όμως λίγο γιατί ε, κατά μέσον όρο περισσότερες από το 70% των δραστηριοτήτων σε αυτόν τον τομέα είναι ε, εφαρμογές λογισμικού σε σχέση με το ICT. Άρα λοιπόν ε, ε, μέσα είμαστε κι εμείς. Η ASD e αντιπροσωπεύει τους τομείς άμυνας ασφάλειας διαστήματος αεροναυτικής από 20 χώρες στην Ευρώπη είναι η φωνή 2.000 εταιριών και 80.000 προμηθευτών, εκ των οποίων πολλοί είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το 2010 ε, αυτό αντιπροσώπευε περισσότερους από 700.000 εργαζομένους και δημιούργησε έναν κύκλο εργασιών περίπου 163 δις ευρώ. Σήμερα θέλουμε να επικεντρωθούμε στους τομείς αεροναυτικής διαστήματος και ασφάλειας που είναι το μη στρατιωτικό κομμάτι των δραστηριοτήτων μας και το οποίο απεδείχθη ότι είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο με τις ευρωπαϊκές στρατηγικές και πολιτικές γιατί εμείς χαιρετίζουμε ε, ως ASD την οριζόντια προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της αντίληψης περί καινοτομίας στο Horizon 2020, γιατί έτσι θα έχουμε άμεση σύνδεση και πιο οργανική συνεργασία μεταξύ των τομέων μας και των ερευνητικών κέντρων και των πανεπιστημίων. Ε, σήμερα θέλω να σας μιλήσω για τις δικές μας απόψεις σε σχέση με το ε, πώς θα γίνει ο προγραμματισμός της έρευνας στην Ευρώπη και θα σας ε, ε, παρουσιάσουμε και την εμπειρία που αποκτήσαμε από την οικοδόμηση της έρευνας στην Ευρώπη. Επειδή είναι κλειδί και καινοτομία, οι κλάδοι μας επενδύουν σε αιτήσια βάση κατά μέσον όρο το 12% των εσόδων τους στην έρευνα και την ανάπτυξη, ούτως ώστε να παρουσιάζουν περιβαλλοντικά φιλικά και λειτουργικά αποτελεσματικά και αποδοτικά προϊόντα στις αυξανόμενες παγκόσμιες αγορές κάτω από σκληρό ανταγωνισμό. Οι κλάδοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να ανταγωνιστούν με βάση την τιμή με τις χώρες BRICS. Πρέπει λοιπόν να κάνουν καινοτομία, τεχνολογία για να διατηρήσουμε τον ανταγωνιστικό διαφοροποιητή της Ευρώπης είναι σημαντικό να διατηρήσουμε τη συνέχεια και την ορατότητα. Για την ε, ε, συνέχεια να δώσω ένα παράδειγμα για να σας δείξω με ε, το ρόλο που παίξαμε στην ευρωπαϊκή έρευνα. Ο κλάδος της αεροναυτικής έχει υψηλή διασύνδεση με τους προμηθευτές ε, μεγάλες επιχειρήσεις ε, στηρίζονται από χιλιάδες προμηθευτές και προμηθευτές προμηθευτών. Είναι μια αλυσίδα αυτή ε, προμηθειών ισχυρή και αξιόπιστη που αποτελείται κυρίως από ΜΜΕ και είναι απαραίτητη για το τομέα μας και πρέπει να θυμόμαστε ότι μας πήρε χρόνια να δημιουργήσουμε και να διατηρήσουμε αυτό το δίκτυο. Οι σχέσεις με τις μικρότερες επιχειρήσεις λοιπόν είναι μάλλον μια εταιρική σχέση παρά μια απλή συνεργασία πελάτη-προμηθευτή. Και εκτός αυτού ήδη έχουμε μια πολύ στενή και μακροχρόνια συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα και τις ερευνητικές ε, οργανώσεις και ιδρύματα. Και έτσι προσπαθούμε να γεφυρώσουμε το κενό μεταξύ της βασικής πρώιμης έρευνας και των πρακτικών εφαρμογών. Σημειώνω επίσης ότι στην κοινότητα των ε, ενδιαφερομένων, εμπλεκομένων έχουμε ε, αεροδρόμια, αεροπορικές εταιρείες, ε, παρόχους υπηρεσιών για την αεροναυπήγηση. Υπάρχει ήδη λοιπόν οριζόντια συνεργασία για να επιτύχουμε τους στόχους του Horizon 2020. Αυτή η κοινότητα στην πραγματικότητα αποτελεί το έργο του ΑΚΑΡΕ, που είναι το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο για την έρευνα στην αεροναυτική στην Ευρώπη, το οποίο ιδρύθηκε περίπου πριν από 12 χρόνια. Επίσης, η τεχνολογική πλατφόρμα ε, υλοποιεί τις ε, κατευθυντήριες γραμμές του Flight Path 2050, και που ε, ε, εγκρίθηκε από τον Αντιπρόεδρο Καλάς και, τον, ε, και την Επίτροπο Τζόγαν Κουίν. Είναι ένα όραμα αυτό για μας με ορίζοντα το 2050. Η προσέγγιση μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, προγραμματισμού που εγκρίθηκε από το ΑΚΑΡΕ ε, έχει να κάνει με τις ιδιαιτερότητες του τομέα της αεροναυπηγικής. Εμείς έχουμε υψηλή έντασης κεφαλαίου και τεχνολογίας προϊόντα, ε, υψηλή συνθετότητας, τα οποία στηρίζονται πολύ στην έρευνα. Η δομή του ΑΚΑΡΕ απεδείχθη πάρα πολύ ε, επιτυχής στο παρελθόν. Έτσι λοιπόν χρησιμοποιείται ως καλό παράδειγμα αυτό το γνωμοδοτικό συμβούλιο και για άλλους τομείς όπως το τομέα της ασφάλειας και του διαστήματος. Ο τομέας του διαστήματος στηρίζει τη δημιουργία παρόμοιας προσέγγισης μέσα από ε, μια ατζέντα στρατηγικής έρευνας που συμπεριλαμβάνει τη βιομηχανία, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις υπηρεσίες του διαστήματος. Το Horizon 2020 θα πρέπει να είναι σημαντική συμβολή σε μια σύντονη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που θα μειώσει την εξάρτηση από μη ευρωπαϊκές πηγές και θα παράσχει πλαίσιο για την ορίμανση των τεχνολογιών του διαστήματος ε, ώστε να περάσουν σε τροχιά πλήρως ε, καταξιωμένες. Ε, επίσης η, στον τομέα της ασφάλειας ε, θα πρέπει να υπάρχει μια ε, πλατφόρμα καινοτομίας ε, για όσους δραστηριοποιούνται στον τομέα της ασφάλειας λαμβάνοντας υπόψη την φωνή της βιομηχανίας. Αυτά τα παραδείγματα δείχνουν την ανάγκη για συνέχεια όλων αυτών των μέσων που πρώτο χρησιμοποιήθηκαν από το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο και θα συνεχιστούν. Έχουμε το παράδειγμα του Clean Sky, καθαρή ουρανή. Αυτό το, αυτή η σύμπραξη ιδιωτικού δημοσίου τομέα είναι παράδειγμα αποτελεσματικής ε, συνεργασίας για την έρευνα μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μεγάλων εταιριών αεροναυτικής, ερευνητικών κέντρων, πανεπιστημίων και πολλών μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και αν θέλουμε να δούμε συγκεκριμένα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυτές ε, είχαν ποσοστό επιτυχίας 40% στους ανοιχτούς διαγωνισμούς σε σύγκριση με 10-15% γενικότερα. Είναι λοιπόν ζωτικό το δίκτυο μεταξύ μεγάλων βιομηχανιών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Όταν δουλεύει αυτό καλά, δίνει μεγάλα ωφέλη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για την ορατότητα χαιρετίζουμε ιδιαίτερα την προσέγγιση της κυρίας Ριέρα Μαντουρέλ όταν ε, λέει και παραθέτω είναι πολύ ευπρόσδεκτη προσθήκη αν η Κομισιόν παρουσιάσει ενδεικτικό καταμερισμό όπου οι πιστώσεις από κάθε μία από τις νομικές βάσεις του Horizon, Horizon 2020 θα ε, διαφοροποιούνται σαφώς τέλος του παραθέματος. Παράλληλα, χαιρετίζουμε και την πρόταση της κυρίας Ριέρα Μαντουρέλ σε σχέση με τον προτινόμενο συνδυασμό θεμάτων ε, κάτω από κοινωνίες ασφαλής και νοτόμους χωρίς ε, αποκλισμούς. Αυτό είναι μια πρόκληση. Το πρόγραμμα θα εξυπηρετηθεί καλύτερα με μια υποδιέρεση μεταξύ κοινωνιών χωρίς αποκλισμούς και καινοτόμους από τη μία πλευρά και ασφαλής από την άλλη. Ε, έτσι ε, δίνουμε περισσότερη έμφαση ταυτόχρονα στην κοινωνική διάσταση της επιστήμης και διασφαλίζουμε σημαντικές εφαρμογές για την κοινωνία όπως διαχείριση των κρίσεων, πολιτική προστασία. Ε, αυτές είναι παρεμβάσεις που χρειάζονται τεχνολογική βελτίωση. Τέλος, να πω κάτι και για ένα θέμα το οποίο ήδη το ανέφερε ο κύριος Έλερα δηλαδή τις προτεραιότητες για τους κανόνες συμμετοχής. Εδώ υπάρχουν τρία θέματα. Η προβλεψιμότητα, η μη διάκριση και η ε, κατάργηση αποκλεισμών. Για την ε, προβλεψιμότητα υπάρχει εδώ μια βεβαιότητα σε σχέση με το ποσοστό χρηματοδότησης. Ο κανόνας του καταμέγιστον 100% δεν βοηθάει τις, ε, τους φορείς να, να, ξέρουν εκείνες τι θα, λεφτά θα βάλουν από την αρχή. Επίση, η μη διακρίση αναφέρεται στην αναγνώριση του πραγματικού κόστου από του διάφορου φορεί όταν συμμετέχουν στα προγράμματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση ένα καταποκοπή ποσό 20% για έμεσο ε, επιλέξιμο κόστος μπορεί να πλουστεύει τα πράγματα αλλά μπορεί να ε, τιμωρεί κάποιους φορείς γιατί ο κανόνας αγνοεί εκείνο το μέρος του κόστους πέρα από το ποσοστό το οποίο είναι απαραίτητο. Τώρα, για το ότι πρέπει να συμπεριλαμβάνονται τα σχετικά ή σημαντικά κόστη, εδώ θέλουμε να παραπέμψουμε στο κόστος διαχείρισης ε, που πρέπει να εντοπιστεί και να καλυφθεί. Τα καλύτερα αποτελέσματα από τα έργα είναι αποτέλεσμα και αποτελεσματικής διαχείρισης και αυτό συνεπάγεται χρήματα. Ε, πολύ σημαντικό είναι και το θέμα των ε, δικαιωμάτων ε, πνευματικής ιδιοκτησίας ε, καλύπτονται από τις ήπα ε, πάρα πολύ αποτελεσματικά. Ε, εδώ η ελεύθερη πρόσβαση στα αποτελέσματα δημιουργεί ένα ρίσκο γιατί χωρίς επαρκή προστασία η έρευνα, η ανάπτυξη και όλες οι σχετικές διαδικασίες καινοτομιών δεν θα ωφελήσουν τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες αλλά θα πάνε αλλού. Τέλος, θέλω να υπογραμμίσω τη σημασία των αποτελεσμάτων που έχουν μέχρι τούδε από κοινού επιτευχθεί. Οι δραστηριότητε έρευνας και ανάπτυξης που έλαβαν χώρα στα πλαίσια των προγραμμάτων ε, πλαίσιο 6 και 7, δραστηριότητες και πρωτοβουλίες όπως το ΣΕΖΑΡ, ένα παράδειγμα παραθέτω μόνο εδώ, επιτρέπουν στην Ευρώπη να παραμείνει ελεύθερη ε, από κανονιστικά, ρυθμιστικά περιβάλλοντα τα οποία ε, θεσπίζονται από πολιτικούς αρμόδιους εκτός Ευρώπης. Επίσης, τα ερευνητικά προγράμματα στην Ευρώπη έχουν την προστιθέμενη αξία και μάλιστα συμβάλλουν σε αυτό να δημιουργήσουν μια πραγματικά ευρωπαϊκή ταυτότητα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Μπερτολόνε και τώρα ο κύριος Γιάν Μέγγελερες, ε, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Έρευνας και Ανάπτυξης, ΕΑΡΤΟ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Έλερα, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι. Για μένα είναι μια μεγάλη τιμή. Να μπορέσω να σας εξηγήσω ε, το έργο το έργο το δικό μας σε σχέση με το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι μεγάλη ημέρα, ήταν μεγάλη μέλη για όλους τους, μέρα για όλους τους συμμετέχοντες. Θα ήθελα να σας αναφέρω ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο φόρουμ καινοτομία και έρευνα στα πανεπιστήμια χαρακτηρίζονται από εξαιρετική ε, βασική έρευνα και σκοπός μας είναι να εφαρμόσουμε την έρευνα αυτή. Μία συχνή παρανόηση είναι ότι η καινοτομία βασίζεται μόνο στην ακαδημαϊκή έρευνα. Οι εφαρμοσμένες ε, έρευνες του ERTO είναι πολύ σημαντικό στοιχείο συμπληρώνουμε τα πανεπιστήμια με την εφαρμογή της έρευνας, μετατρέποντας ε, τις ανακαλύψεις σε εφαρμόσιμη τεχνολογία που θα μπορέσουν να τα χρησιμοποιήσουν όσο πιο πολλοί χρήστες γίνεται. Τα πανεπιστήμια ε, έχουν την αριστεία, αν θέλετε, την επιστημονική. Εμείς έχουμε την επιστημονική συνάφεια όμως. Χρειαζόμαστε και προωθούμε τη συνεργασία με τα πανεπιστήμια και με μεγάλες ε, επιχειρήσεις. Είναι, είμαστε η Ευρωπαϊκή Ένωση για Οργανισμούς Έρευνα και Τεχνολογίας. 150, 350 ε, επιχειρήσεις ε, εκπροσωπούμε. Μία έρευνα του 2011 καταδεικνύει 150 ερευνητές, 100.000 ε, πελάτες και μεγάλη αξία η οποία έχει γεννηθεί τα τελευταία χρόνια. Έχουμε 25% του προγράμματος πλαισίου. Και από ό,τι ξέρουμε το έκτο πρόγραμμα, δηλαδή ξέρουμε ότι έχουμε το 35% το, το οποίο εισφέρεται όσον αφορά αυτού του συνεργαστέ. Και επίση θα πρέπει τώρα να σκεφτούμε ότι έχουμε μια τέτοια συστήματα τα οποία να μην γνωρίζουν σύνορα. Θα πρέπει να σκεφτούμε ότι έχουμε την δύναμη τη χειροτομία, ώστε να μπορέσουμε να, να βελτιώσουμε τη ζωή των Ευρωπαίων και θα πρέπει να ε, προχωρήσουμε σε, σε εφευρέσεις, σε καινοτομία, σε, σε, σε αξιοποίηση. Οπότε θα πρέπει η γνώση να βοηθήσει την βιομηχανία για τους τρόφους και οπότε αυτό μας το, το, το δίκτυο είναι ένας καταλήτης θετικός για την εξέλιξη και για τις ΜΜΕ και για τις ε, πολυεθνικές, ούτως ώστε να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη προσβασιμότητα. Και όπως ε, φάνηκε από το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο, η συνεργασία αυτή αφορά ε, τους βασικούς συντελεστές οι οποίοι μπορούν να, να δώσουν το κίνητρο για την αλυσίδα της ε, Και έτσι μπορούμε να τονίσουμε ε, την ανταγωνιστικότητα και έτσι μπορεί όλη η κοινωνία να ωφεληθεί. Οπότε έχουμε αυτή μια τέτοια ανάλυση από τα, τα μέλη μας για το 7ο πρόγραμμα έδειξε ότι ε, ε, μόνο αυτών των, των συντηρητικών μας συντελεστών εισφορά ήταν όσο όλων των άλλων και επίσης και οι ΜΜΕ συμμετέχουν πάρα πολύ και ως ε, ε, πρόεδρος του, του, του, του φορέα αυτού για την, ε, για την έρευνα ε, θέλω να σας πω ότι δίνουμε μεγάλη σημασία όσον αφορά την καινοτομία και έχουμε αυτό, αυτή την διάρθρωση των τριών πυλώνων οπότε μπορούμε να έχουμε ε, μακρόπνοη προγραμματισμό και σε καινοτομία μεσοπρόθεσμη και βραχυπρόθεσμη μπορούν να μας οδηγήσουν σε πρωτοπορία στον τομέα της βιομηχανίας. Όσον αφορά τον πρώτο πυλώνα, η αριστεία, η επιστημονική είναι κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει και υποστηρίζουμε την έρευνα γιατί θέλουμε να γίνει μια επανεξισορρόπηση του, του, του, του σχετικού προϋπολογισμού για τις αναδυόμενες τεχνολογίες και θα πρέπει να στοχεύσουμε όσον αφορά τις, ε, τους στόχους για την πρωτοπορία στη μηχανία και τους στόχους για την κοινωνία επίσης, τις προκλήσεις. Επίσης ε, θα πρέπει να υπάρχει ε, φροντίδα για τις υποδομές και το ότι δίνουμε για αυτές τις κοινωνικές αλλαγές, για τις προκλήσεις θα μας βοηθήσουν να πετύχουμε τους στόχους της πολιτικής του 2020 και μεγάλη μας χαρά βλέπουμε ότι δίνεται ιδιαίτερη έμφαση ε, στα μέσα επίτευξης αυτής της πρωτοπορίας με, ε, με, με την τεχνολογία. Χρειάζεται επομένως να δούμε πώς με τον καλύτερο τρόπο θα εφαρμόσουμε αυτά τα οποία έχουν αποφασιστεί. Από πολλές απόψεις, οι, οι κανόνες συμμετοχής για τον 2020 αντικατοπτρίζουν τους κανόνες του 7ου προγράμματος πλαισίου ε, και υπάρχει ένα στοιχείο συνέχεια και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να απλουστεύσει το πρόγραμμα ούτω ώστε να ωφεληθούν ε, οι επιλέξιμοι όμως θα πρέπει να μην θίγονται άλλοι εμπλεκόμενοι. Το πιο σημαντικό εδώ είναι το, το, μοντέλο της χρηματοδότησης που αφορά το, το, αφορά το τι προβλέπεται όσον αφορά τον ε, ρυθμό ε, χρηματοδότηση και συγχρηματοδότηση. Σύμφωνα με αυτό το, το, το πρόγραμμα 75% ήταν η χρηματοδότηση που δόθηκε. Σύμφωνα με το Horizon 2020 έχουμε, έναν, ε, θα έχουμε 60% χρηματοδότηση. Είναι απλά οικονομικά. Ποιος θα, και απλά μαθηματικά ποιο θα πληρώσει το υπόλοιπο 40%. Ο προτινόμενο κανόνας του άρθρου 22 λέει ότι η εισφορά των, των, τρίτων δεν πρόκειται να μετρήσουν ως ε, κόστη επιλέξιμο. επομένω, το υπόλοιπο 40% θα προέλθει από εσωτερικούς πόρους. Επομένω, το πρόγραμμα είναι ότι οι περισσότεροι ερευνητέ δεν έχουν τέτοιου πόρου. Επομένω. αυτό σημαίνει ότι οι συμμετέχοντες πρόκειται να αναγκαστούν να μειώσουν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Έγινε μια έρευνα από το φορέα μας που λέει ότι οι μισοί πρόκειται να μειώσουν τουλάχιστον 20% τη συμμετοχή τους. Επίσης, οι άλλοι μισοί πρόκειται να δώσουν υπολογιστή. Και έχουμε τώρα τους, τους κανόνες για το 2020 που επί χρόνια έχει ενθαρρύνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτοί που συμμετέχουν στα προγράμματα να, ε, να, να, να, κινηθούν προς, μια ε, υποχρέωση λογοδοσίας τόσο ώστε να υπάρχουν ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των ε, διαφορετικών εμπλεκομένων στην έρευνα. Οπότε ε, όσον αφορά το έμεσο κόστος πάμε προς τα πίσω και έχουμε αυτό το ποσό το σταθερό και αυτό θα, αν θα καλύψει ε, τόσα πολλά πανεπιστήμια που θέλουν να συμμετέχουν στο, στο πρόγραμμα και επομένω έχουν πει πολλά πανεπιστήμια ότι πρόκειται για πιστοδρόμη σε σχέση με το ευρώ πρόγραμμα πλούσια, γιατί είναι αυτό αρνητικό σήμα, αρνητικό μήνυμα προς τα πανεπιστήμια και προς τις ε, αρχές όσον αφορά ε, τι μεθοδολογίε και όσον αφορά το, το, το, τον τρόπο χρηματοδότηση σε σχέση με το, το σταθερό ποσό. Από 35 χώρες προέρχεται αυτή η συμμετοχή και λένε αυτοί ότι αυτού του είδους τα λογιστικά πρότυπα πρόκειται να οδηγήσουν σε ε, θα οδηγήσουν σε τέτοιο καθεστώς που δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό. Υπάρχει μια επιλογή όσον αφορά τα άμεσα κόστη σε σχέση με αυτό που ήσχαν στο 7ο πρόγραμμα. Ε, θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σωστά να κάνει απλουστεύσει και επομένω μια τέτοια αναλλακτική, α πούμε το 75% ε, της, ε, της επιστροφής εξόδων να αφορά το έμεσο κόστο και το 75% σαν ένα σταθερό ποσό συμμετοχής για αυτά τα κόστη. Εμείς θεωρούμε ότι οι περισσότεροι ερευνητές ε, επιλέξιμοι θα το, θα το δεχθούν. Οπότε θα πρέπει να υπάρχει μια τέτοια επιλογή, τουλάχιστον για του μη κερδοσκοπικού οργανισμού έρευνα να μπορούν να ζητήσουν επιστροφή του, το το το έμεσου κόστου. Και εάν επιμένει οπωσδήποτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μείνει σημερινή το μοντέλο του 100% 20% αυτό θα το δεχτούν οι ερευνητέ ε, και να υπάρχει η επιλογή τα, οι μη κερδοσκοπικέ οργανώσει να μπορέσουν να μπορούν να ζητήσουν το εξόδια. Τώρα θέλω επίση με το λίγο χρόνο που έχω να σα επισύρω την προσοχή σε άλλε δύο πτυχέ των όσων ε, προτείνονται για τη συμμετοχή. Το Horizon 2020 αφορά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα το οποίο προτείνεται. Όμω, από ό,τι φαίνεται, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, λέει να υπάρχουν ε, διαφορετικές ρυθμίσει ανάλογα με την κάθε δράση, τον κάθε στόχο και σε μερικέ περιπτώσει να φτάνει στο το 70% στην χρηματοδότηση. Αυτό δεν πρόκειται να δεν να, να, να, να φέρει κοντά την έρευνα με την καινοτομία, θα τις απομακρύνει. Και έτσι θα χάσουμε έδαφος μήνες αν όχι χρόνια. Τα δεδομένα, οι στόχοι της έρευνας όπως τίθενται είναι πάρα πολύ αξιόλογοι, αλλά θα πρέπει να δούμε ήδη τώρα τι ανήκει στο, στο, στο δημόσιο τομέα. Χρειάζεται να, υπάρχει, να είναι εφαρμόσιμο όσο προβλέπονται και άρα δεν θα πρέπει να αποθαρρύνουμε τους ερευνητές και θα πρέπει τα δεδομένα να είναι προσβάσιμα σε όλους. Το ορίζον 2020 είναι άριστο πρόγραμμα. Τα υπέρ του είναι η απλούστευση των διαδικασιών, τον φέρουμε κοντά καινοτομία και έρευνα, το, οι προκλήσεις για την κοινωνία, η ΜΜΕ, περισσότερη προσπάθεια, όλα αυτά είναι θετικά. Όμως θα πρέπει να προσέξετε τον ρόλο αυτών των, ε, των, των φορέων και επίσης πολύ βασικό είναι το, αυτού του είδους το προτινόμενο μοντέλο χρηματοδότηση που θα, απο, αποθαρρύνει πάρα πολλούς ε, πολλά μέλη του, του φορέα μας. Grazie. La parola per l'ultimo είναι η τελευταία που θα λάβει το, τον λόγο. Είναι αντιπρόεδρος ε, του, του Ιδρύματος ε, Στρατηγικής του Πανεπιστημίου του Cambridge. Πρόεδρε, κύριε Έλλερ, καλωσορίζουμε την ευκαιρία που μας δίδεται να παρουσιάσουμε τα στοιχεία μας. Θα ήθελα στο τέλος της ημέρας να δώσω μία προσεκτική νότα αισιοδοξία, γιατί προέρχομαι από ένα τομέα που έχει πολλές από τις λύσεις των προβλημάτων που συζητάμε σήμερα, αλλά πριν ξεκινήσω θα ήθελα να πω ότι ο συνάδελφος από την ΙΑΡΤΟ ανέφερε θέματα απλοποίηση με τέτοιο καλό τρόπο που δεν θα το αναφέρω εγώ στη δική μου παρουσίαση γιατί ανέφερε πολύ καλύτερα τα όσα ήθελα να πω εγώ και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Ήθελα να θέσω δύο, τρία ερωτήματα προς την αίθουσα. Γιατί χρειάζονται προτεραιότητε ε, στο πρόγραμμα ε, ορίζοντας 2020, γιατί έχει σημασία η αριστεία και πώς το πρόγραμμα ορίζον 2020 μπορεί να ωφελήσει όλη την Ευρώπη, γιατί εκπροσωπώ 24, 24 από τα πιο υψηλού κύρους πανεπιστήμια στον κόσμο και θα ήθελα να συζητήσουμε πώς ε, τα ωφέλη θα αγγίξουν όλα, όλες τις χώρες και όχι μόνο τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ευρώπη, Καταλαβαίνω τη διάκριση μεταξύ έρευνας ε, και καινοτομίας. Δεν νομίζω ότι αυτό αποτέλεσε ιδιαίτερα θέμα τα τελευταία 20 χρόνια όταν ξεκίνησε η εξωτερική ανάθεση της έρευνας και της ανάπτυξης σε μεγάλα πανεπιστήμια στον κόσμο. Δεν είναι ασυνήθιστο να βρω ένα συνάδελφο ο οποίος έχει βγάλει εκατομμύρια από ένα σπίνα ότι δεν μπορώ να δυσκολευτώ να φανταστώ μια βασική επιστημονική ανακάλυψη να οδηγήσει σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά νομίζω ότι αυτό αποτυπώνεται πολύ καλά στο πρόγραμμα Horizon 2020, ότι πρόκειται για ένα σύστημα όπου τα πανεπιστήμια παίζουν έναν κρίσιμο ρόλο. Δεν είμαι συνηθισμένη σε προγράμματα πολιτικής ε, που μου με ενθουσιάζουν, αλλά με ενθουσίασε το πρόγραμμα αυτό. Μιλάει για καινοτομίες από νέες τεχνολογίες, από αναδυόμενες τεχνολογίες και το πρόγραμμα Horizon 2020 θα επιτρέψει στα πιο λαμπρά μυαλά να ενισχύοντας μάλλον δραστηριότητες όπως το ERC, το Marie Curie και συγκεκριμένα εργαλεία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το σημαντικό είναι ότι περιγράφει ένα σύστημα δεν πρόκειται για χαοτικούς παράγοντες που με καυκαϊκό τρόπο εργάζονται. Όχι, πρόκειται για συγκεκριμένα τμήματα της αλυσίδας προμήθειας και που παίζουν σημαντικό ρόλο τα πανεπιστήμια και η έρευνα. Γιατί έχει τόσο μεγάλη σημασία η αριστεία. Στην Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μιλάμε ιδιαίτερα για ε, value for money. Αλλά ένας ομιλητής ρώτησε για τις ε, δημιουργικές βιομηχανίες και είπε ότι θα πρέπει να εστιαστούμε και για, σε θέματα χρημάτων υπέρ των αξιών, money for values, να βρούμε ένα σύστημα για να μπορέσουν να συμμετάσχουν και να συνεργαστούν οι επιστήμονες με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό το οικοσύστημα ακριβώς δημιουργείται. Θα ακούτε ότι μιλάω με αμερικανική προφορά και δεν θεωρώ, επειδή εργάζομαι τα τελευταία, τις τελευταίες τρεις δεκαετίες στην Αμερική, ότι είμαστε πίσω από την Αμερική. Θεωρώ ότι είναι εξαιρετικό το έργο σε ό,τι αφορά την καινοτομία και τη δημιουργικότητα στην Ευρώπη. Και ένα σύστημα που θα προωθήσει όλα αυτά θα κάνει τις ΙΠΑ να κάτσουν και να κοιτάξουν τι κάνουμε. Τέλος, πώς μπορεί το πρόγραμμα να ωφελήσει όλους τους Ευρωπαίους. Θα ήθελα να σας πω ότι στο Πανεπιστήμιο του Cambridge είχαμε φοιτητές από την Τσεχική, Πολωνική και άλλες κυβερνήσεις ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποιος, ε, κάποια από τις ε, φοιτήτριες τη ρώτησα αν ε, θεωρούσε α, επειδή φοιτούσε στο τμήμα μηχανικής τη ρώτησα αν θεωρήσει ότι ήταν δύσκολο το πρόγραμμα και μου απάντησε ότι όχι, τη διασκέδαζε ιδιαίτερα γιατί ξέρετε είναι πάρα πολύ δύσκολο έχει φήμη ότι είναι πολύ δύσκολο το τμήμα μηχανικής μου απάντησε ότι όχι αλλά της λείπει το σπίτι της. Ε, τώρα είναι στο MIT και θα επανέλθει στην Αμερική. Ακριβώς αυτού το τύπου φοιτήτρια θέλουμε να προωθήσουμε με τις δράσεις Marie Curie. Θα συνεχίσει το καθημαϊκό της έργο, αλλά τελικά αυτό που θέλει να κάνει είναι να επιστρέψει στη Ρουμανία και εκεί θέλει να δημιουργήσει, να ιδρύσει μια μικρομεσαία επιχείρηση. Και όταν θα την έχει δημιουργήσει την επιχείρηση αυτή, θα έρθει σε επαφή με συναδέλφους που μπορεί να εξακολουθούν να είναι στο Cambridge για να αντιμετωπίσει διάφορες προκλήσεις. Αν ακούγουμε αν θέλετε, Ευαγγελική, είναι επειδή μεγάλωσα στην Ινδιάνα, που δεν ξέρουν οι πιο πολλοί Αμερικανοί που είναι, να σας διαβεβαιώσω ότι δεν ήταν πολύ ισχυρό το πανεπιστημιακό σύστημα της Ινδιάνα. Υπονομεύτηκε μάλιστα το σύστημα αυτό. Μετά το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο όμως η Ινδιάνα ξεκίνησε με τα πρώτα πανεπιστήμια και προσέλαβε μόνο Ευρωπαίους για να δημιουργήσουν μία από τις καλύτερες ιατρικές, νομικές σχολές αλλά και μουσικά, μουσικές σχολές. Και πάλι στη μέση του πουθενά είναι οι σχολές αυτές, αλλά καταδεικνύει το παράδειγμα αυτό ότι ένα πρόγραμμα όπως το Horizon 2020 δημιουργούν, δημιουργεί ευκαιρίες για κράτη-μέλη που ελπίζουν σε τέτοιες ευκαιρίες. Εδώ εκπροσωπώ σήμερα την ομάδα Russell και είμαστε έτοιμοι να διαδραματίσουμε το ρόλο μας στο πρόγραμμα αυτό. Δεν είναι υποτιμούμε τις δυσκολίες, αλλά θεωρούμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλο δυναμικό στην Ευρώπη που μπορεί να ανταποκριθεί στα προβλήματα αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Βανίστελ Ρόι. Thank you, thank you very much ευχαριστώ. Ήταν ε, μακριά η ημέρα για όλους μας. Υπάρχει πρόγραμμα ανταλλαγών και για ερευνητέ και βοηθούς πανεπιστημίων σε όλη την Ευρώπη, ε, το οποίο το προωθεί η Επιτροπή Ήτρε. Κάναμε τις ανταλλαγές αυτές και έχετε και δίκιο για την αριστεία που έχουμε και έχουμε καλά αποτελέσματα έτσι. Το πρόβλημά μας δεν είναι εκεί. Το πρόβλημα είναι να πάμε μέχρι την αγορά. Δηλαδή να συνεχιστεί η αλυσίδα της καινοτομίας, όπως είπε και ο εκπρόσωπος των ERTOs. Η ερώτηση λοιπόν είναι, ποια μέσα μας λείπουν, αν δούμε και τους κανόνες συμμετοχής, αν δούμε τη βιομηχανία, βλέπουμε, ας πούμε, οι βασικές διευκολυντικές ε, τεχνολογίες και πρωτοβουλίες. Συνήθως όλα αυτά τα πράγματα όταν καταλήξουν στην, σε νέες αλυσίδες παραγωγής φεύγουν από την Ευρώπη και πάνε σε άλλα μέρη του κόσμου για να γίνει αυτό το κομμάτι. Εμείς τι θα κάνουμε για να κρατήσουμε αυτό το κομμάτι. Γιατί αυτή η αλυσίδα υψηλής αξίας πρέπει να μείνει εδώ, με καινούργια κίνητρα, τις βασικές διευκολυντικές τεχνολογίες, τις μελλοντικές βιομηχανίες, να έχουμε καλύτερα προγράμματα κατατικών ενισχύσεων. Τι να κάνουμε, μπορείτε να μας πείτε εσείς. Ναι, σύντομα να απαντήσω, αλλά φαντάζομαι θα συμπληρώσουν και οι συνάδελφοι. Α, ο κύριος Γκλάντε. Πρώτα ερωτήσει. Ναι, έχουμε σκληρούς κανόνες εμείς εδώ. Δύο ερωτήσεις. Μίλησα και στο Εδιμβούργο λίγες μέρες πριν. Ε, πρόκειται αυτό γιατί το διπλό σύστημα για την υποβολή των προτάσεων. Κάποιοι είπαν ότι καλό είναι, δεν ολοκληρώνουμε το, τη διαδικασία με την πρώτη πρόταση. Είναι υπέρ της διπλής προσέγγισης. Άλλοι λένε, μα τόσο πολλή δουλειά να κάνουμε ε, αν δεν κάνουμε πάρα πολλή δουλειά θα υποληφθούμε στην αξιολόγηση ε, οπότε είναι κατά του διπλού συστήματος υποβολής εκθέσεων καλό είναι ή κακό επίσης ο κύριος Μπερτολόνε μίλησε για τις πατέντες, τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας κλπ θα ήταν χρήσιμο να βάζαμε ότι πρέπει εκ των προτέρων να υπάρχει συμφωνία για το ποιο θα, χρησιμοποιηθεί, θα χρησιμοποιεί τα διπλώματα ευρεσιτεχνία και τι προσέγγιση θα ακολουθηθεί. Γιατί είναι λίγο γενικόλογο το σχετικό εδάφιο. Δηλαδή, αφού ολοκληρωθεί κάποιο αποτέλεσμα, δεν είναι σαφές σε ποιον θα ανήκει το, η, η πατέντα, η ευρεσιτεχνία. ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όσον αφορά την ε, απλούστευση. Το Λόγο Κοινοβούλιο έχει βρει κάποιο είδου ε, τέτοια πλειοψηφία, ώστε να μπορεί να καλύψει ε, το αίτημα της απλούστευσης από πλευράς των επιλέξουμε και συμφωνώ με αυτό, αυτά τα οποία ακούσαμε και κυρίως με τον ε, πρόεδρο της ΕΡΤΟ ότι όσον αφορά αυτές τις ε, πολιτικές πλειοψηφίες έχουμε συμπαραταχθεί και έχουμε πει από την μεριά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν ξέρω μήπως θα πρέπει να υπάρξει μια τέτοια πρωτοβουλία συνεννόηση μεταξύ των υπηρεσιών που ασχολούνται με την έρευνα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με φορεία γίνονται που ασχολούνται με τα οικονομικά. Διότι αναφέρεται στο έγγραφο ότι υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία ε, καλύπτονται για στην τριετή αναθεώρηση ε, του δημοσιονομικού κανονισμού. Νομίζω όμω ότι όσον αφορά το Κοινοβούλιο θα πρέπει να ληφθεί μια τέτοια πρωτοβουλία. Τελευταία παρατήρηση τώρα όσον αφορά τη συμμετοχή και κυρίω όσον αφορά ε, ε, την πρόκληση που ονομάζεται ευφυής, μεταφορά κλπ. Νομίζω ότι θα πρέπει αυτό να καλύψει όσο είναι περισσότερους τομείς, γιατί αναφέρεται εδώ η, αεροπορία, η αεροπλοεία, οι αερομεταφορές και οπότε θα, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι πρόκειται για, για κάποιους τομείς έντασης τεχνολογίας. Άρα θα πρέπει να έχουμε, εδώ θα έχουμε ανταγωνισμό με όλο τον πλανήτη και άρα θα πρέπει η τεχνολογία να είναι προηγμένη όσον αφορά τις προηγούμενες γενιές αεροσκαφών και άρα αυτό θα πρέπει να αναφέρεται όσον αφορά την, ε, το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν ξέρω τι πρεσβεύει το πάνελ σε σχέση με αυτό. Ο κύριος Κέλλη. Μακρά η μέρα, αλλά αξιόλογη γιατί είχαμε όλα αυτά τα οποία μάθαμε και ακούσαμε. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει, αν εφαρμοστούν όλα αυτά, ναι, θα γίνει πιο ε, πιο ανταγωνιστική Ευρώπη. Υπάρχει κάτι το οποίο με προβλημάτισε. Αυτό που είπε ο κύριο Μάγκης. Όσον αφορά τις αλλαγές στη χρηματοδότηση από 75% θα πάει στο 60%. Και έτσι αντί να έχουμε περισσότερη έργο θα έχουμε λιγότερη. Για πέστε μας περισσότερα για να δούμε τι θα πρέπει να γίνει. Αλλά επίσης να, να, σχολιάσει και η Επιτροπή πάνω σε αυτό. Γιατί είναι απίστευτο μία πρόταση που έχει ως στόχο την αύξηση της έρευνας και τον έννοι έρευνα πιο εφαρμόσιμη να έχει τα αντίθετα αποτελέσματα στην πράξη. Signora Κυρία Φόρτ, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, Δόκτωρα Πάντς για την ε, έμπνευση που μας έδωσε στο τέλος της ημέρας. Γιατί το Cambridge ε, είναι έμπνευση όχι μόνο ως πανεπιστημίο, αλλά και ως κλάστερ για μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί. Συχνά μιλάμε για clusters ως τμήμα της επόμενης φιλοδοξίας μας. Αλλά θα μιλάτε στους φοιτητές σα σήμερα, στο παράδειγμα που μας δώσατε, η φοιτητριά σας θα ήθελε να υπάρχει ένα τέτοιο κλάστερ ή θα ήθελε να δουλεύει σε ένα εικονικό κλάστερ, δηλαδή να επιστρέψει στη Ρουμανία και να συνεργάζεται με τους ε, συμφοιτητές της, με τους συνεργάτες της. Άρα, μήπως πολλά από αυτά θα μπορούσαν να γίνουν για την επόμενη γενιά σε εικονικό επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ένα λεπτό για τις απαντήσεις. Δυστυχώς είναι κάπως περίεργο αυτό, αλλά δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πρώτη ερώτηση. Να αναφέρω μία δυνατότητα δύο δυνατότητε. Η μία περιγράφεται στο πρόγραμμα Horizon 2020 το γεγονός ότι θα πρέπει να εξετάσουμε την παραγωγή ως ε, υψηλής τεχνολογίας δραστηριότητα με τον όρο ότι θα παραμείνουμε ανταγωνιστικοί και στην ε, παραγωγή. Δεύτερο σημείο. Θα πρέπει σε κάποιες περιπτώσεις να υποκινήσουμε και να διοχετεύσουμε τις ε, προσπάθειες στα πλαίσια του PMI. Σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και πανεπιστημίων προ όφελο μια καλή ε, μικρή επιχειρήση για το IPR. Νομίζω ότι επιλύσαμε το θέμα με το IPR όταν τελικά θέσαμε το θέμα των διπλωμάτων ευρεσιτεχνία. Αν είμαστε ισχυροί στο θέμα των ευρεσιτεχνιών, θα είμαστε ισχυροί και στην αγορά των ευρεσιτεχνιών και τότε θα αντιμετωπίσουμε το θέμα του IPR. Σύμφωνα απολύτως για το γεγονός ότι τα κλάστερ, ό,τι όνομα και να τους δώσουμε, αποτελούν σημαντικό τμήμα του οικοδομήματος για τις οριζόντιες δραστηριότητες που ορίζονται στο ορίζον 2020. Ε, Ο κύριος Μέγκελερς. Λόγω του προχωρημένου χρόνου, εγώ θα απαντήσω σε δύο ερωτήσεις των κυρίων Κέλλη και Βανίστελ Ρόι. Κύριε Κέλλη, αυτό που προσπάθησα να πω είναι ότι γίνεται πολύ έρευνα και υπάρχει πολύ ερευνητικό δυναμικό στο, στην Ευρώπη, στα πλαίσια των ε, προγραμμάτων πλαίσιο. Και με το νέο μοντέλο μπορεί να υπάρξει οπισθοχώρηση. Οι κανόνες μπορούν να βελτιωθούν. Εγώ εξακολουθώ να είμαι υπέρ της απλοποίησης, αλλά θέλουμε και οι RPOs να συμμετέχουν μέσα από την απλοποίηση όλα τα ιδρύματα που ήθελαν σύστημα πλήρους κόστους ε, δεν πρέπει να τιμωρηθούν επειδή είναι διαφανή και το, το πραγματικό έμεσο κόστος να μην την υπόψη. Αυτή είναι η πρότασή μας. Κύριε Βανίστελ Ρόι, αν ε, είχαμε λύσει πανάκια, ή μάλλον αν είχαμε μια ιδεώδη λύση, θα τη λέγαμε. Στην Ευρώπη πάντως ε, έχουμε μεγάλο δυναμικό στις ε, επιστημονικές ε, ε, δραστηριοποιη... δράσεις και σε επίπεδο παραγωγής επίσης. Δηλαδή έχουμε δύο αλυσίδες στην επιστήμη και την παραγωγή που έχουν πλήρως αναπτυχθεί στην Ευρώπη σχεδόν σε όλες τις χώρες. Πρέπει να φροντίσουμε λοιπόν να συντομεύσουμε λίγο αυτές τις αλυσίδες και αν βρούμε λύσεις, και τελειώνω εδώ, Καμιά φορά οι κρατικέ ενισχύσεις θα πρέπει ίσως να ειδωθούν με διαφορετικό τρόπο από ό,τι κάναμε μέχρι τώρα. Ευχαριστώ και η κυρία Τζένιφερ Μπάρνς για να απαντήσω στην πρώτη ερώτηση. Απαντήσατε ήδη. Ε, κάτι άλλο που μένει, είναι λίγο δυσάρεστο, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να το δούμε. Δηλαδή η γραφειοκρατία. Αν είναι το χέρι της βαρύ στο σύστημα, και το συζητήσαμε αυτό, τότε οι ερευνητές στα πανεπιστήμια θα πάνε και που είναι τα περισσότερα χρήματα. Νομίζω ότι υπάρχει επιθυμία να συμβάλλουν στην ευρωπαϊκή ατζέντα, αλλά άμα τους δυσκολέψουν πολύ τη ζωή, θα δυσκολευτούν και αυτοί να το κάνουν η ερώτηση της Βίκη Φόρντ για το φυσικό και το εικονικό. Είναι πολύ ωραία ερώτηση, δεν το είχα σκεφτεί. Ε, σύντομα όμως θα ήθελα να αναφερθώ σε εργασίες που έγιναν στο Cambridge για τις νευροεπιστήμες. Τα εικονικά συστήματα είναι καλά για τον κόσμο, ε, αλλά υπάρχουν και περιορισμοί γενικότεροι σε σχέση με το πώς ε, αλληλεπιδρούμε ε, μεταξύ μας. Είναι ε, πολλές φορές δύσκολο να αντιμετωπίσουμε με εικονικά μοντέλα πραγματικές προκλήσεις. Εκείνο που μπορεί να γίνει όμως είναι να αναμειγνύονται πολύ καλύτερα στο μέλλον τα ε, ε ιδεατά ή τα εικονικά με τα πραγματικά στοιχεία. Ευχαριστούμε κυρία Τζένιφερ Μπάρνς, ευχαριστούμε και τους ε, διερμηνείς. Δεν ξέρω αν μπορούμε να ζητήσουμε λίγα λεπτά ακόμη ούτως ώστε ο Κρίστιαν Έλερ να παρουσιάσει τα συμπεράσματα. Τρία λεπτά για τον Κρίστιαν. Ευχαριστώ. Στο τέλος λοιπόν να μιλήσω στα αγγλικά να κάνω μια σύνοψη. Χαίρομαι που η κυρία Μπάρνς αναφέρθηκε ότι υπάρχουν μεγάλες ευκαιρίες σήμερα για παράδειγμα βάσει του μοντέλου Stanford. Θεωρώ ότι υπάρχει μία ευκαιρία που ύπταται στον αέρα στην παρούσα φάση και νομίζω ότι η πρόταση είναι πάρα πολύ καλή. Γιατί πολλά μπορούμε να πετύχουμε και πολλά έχουμε πετύχει. Και αυτό το θέμα δεν ε, έχει να κάνει μόνο με την ακρόαση. Έχουμε μία μόνιμη ομάδα εργασία. Συμμετείχαμε στη σχετική ομάδα εργασία των Βρυξελών πριν από δύο χρόνια. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Ναι. Νομίζω ότι τελικά αποζητούμε μία λύση opt-out για τα RTOs, αλλά να μην ε, το παρακάνουμε με την απλοποίηση. Είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν λύσεις θα πρέπει να εξετάσουμε το μοντέλο μικτού κόστους. Θα πρέπει να υπάρχει μια πιο συνεκτική ιδέα για το πώς θα εργαστούμε με τα μεικτά μοντέλα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Κοιτώντας την αλυσίδα της καινοτομία από τα RTDs μέχρι την καινοτομία, δεν μπορούμε να έχουμε διαφορετικούς στο μεταξύ, χρειαζόμαστε σε πρακτικούς όρους μοντέλα μεικτού κόστους. Αυτό που θα αποτελούσε τη μεγαλύτερη σύμβολη του Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι η Επιτροπή φοβάται το ελεκτικό συνέδριο και το ελεκτικό συνέδριο έχει πολύ σημαντικό ρόλο να διδραματίσει, αλλά πρακτικά όλα αυτά εξυπηρετούν την ελεγκτική εξουσία του Κοινοβουλίου. Άρα, καλέσαμε και τους ελεγκτές σε θέματα προϋπολογισμού. Άρα, συζητήσαμε με το ελεγκτικό συνέδριο για το τι θα μπορούσε να επιτραπεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κρατώντας την ιδέα ότι είμαστε υποχρεωμένοι να προσπίσουμε το συμφέρον του Ευρωπαίου φορολογούμενου. Νομίζω όμως ότι υπάρχουν ευκαιρίες για την εξέβρεση λύσης. Το Κοινοβούλιο μπορεί να βρει λύσεις για να απαλύνει τον έλεγχο σε θέματα χρηματοδότησης και παράλληλα να αντιμετωπίσει αυτή την ε, μεγάλη πρόκληση της απλοποίησης. Νομίζω ότι τελικά υπάρχει θετικό βήμα θετικό μήνυμα. Έχουμε δουλειά να κάνουμε, την οποία και είμαστε διτεθειμένοι να την κάνουμε. Και νομίζω ότι στην τελική ανάλυση θα δούμε μία απλοποίηση. Και αυτό θα το αισθανθούν και τα εθνικά κράτη-μέλη που θεωρούν ότι υπάρχει ίσω αντιπαλότητα μεταξύ των ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρο για τα μέλη της Επιτροπής Βιομηχανίας. Θα τα πούμε αύριο στις 9.